Chers collègues, je vous invite à prendre place. Αγαπητοί συναδελφοί, σας παρακαλώ να καθίστε. Με μια κάποια καθυστέρηση, για να μην πω και σημαντική, θα ξεκινήσουμε σε λίγα λεπτά. Chers membres, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη αυτή ημέρα της Ολομέλειάς μας που ξέρετε ότι θα συνεχιστεί και το απόγευμα. Και θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που έγινε χτες, τη απουσία μου. Μάρκο, σε ευχαριστώ πολύ, καθοδήγησες με μεγάλη επιτυχία, αν και μεταξύ το ξέρεις το το θέμα, μπορείς να το κάνεις. Ε, καθοδήγησες λοιπόν επάξια της ε, εργασίες με την υιοθέτηση τελικά της, ε, του ψηφίσματος για, την, ε, για τις προοπτικές επιτροπής. Ξέρετε ότι δεν μπόρεσα να έρθω διότι εχθές ήμουνα σε μια εκδήλωση σημαντική που συνοργανώσαμε στις πόλεις του Άχεν, του Μάστριχτ και της Λιέγης μαζί με, την, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πρέπει να πω ότι ήταν εξαιρετικά ε, επιτυχής και αυτή η εκδήλωση. Μου επέτρεψε μάλιστα για άλλη μια φορά να διαπιστώσω το συγκεκριμένο αντίκτυπο που έχει η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών αν φερειπίν τους συμβεί κάτι και έχουν ένα πρόβλημα υγείας σε μια χώρα, σε μια πόλη άλλη από αυτή που ζουν. Η χθεσινή μας απόφαση με το ψήφισμα ήταν και ένα σημείο καμπή σε σχέση μας με τα ε, λοιπά ευρωπαϊκά όργανα. Με το προσχέδιο αυτό, το blueprint που υιοθετήσαμε εν ώψη του στρατηγικού θεματολογίου του Συμβουλίου, που λάβατε πιστεύω όλοι, αλλά και με το ψήφισμα που υιοθετήσαμε χθε. Αποστήλαμε, πιστεύω, ένα μήνυμα περίφραστο, ένα μήνυμα το οποίο θα μετρήσει στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον, χάρη στο οποίο μπορέσαμε και να υπενθυμίσουμε τις θέσεις μας και θα μπορέσουμε να το πράξουμε και στο μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, και πριν κηρύξω πριν αρχίσουμε τι ουσιαστικέ εργασίε μα, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστώ θερμά το γενικό μα γραμματέα, το Γύρι Μπουργιάνεκ, του οποίου η θητεία λύγει σύντομα στι 31 Ιουλίου. Και άρα είναι ε, ευκαιρία για μας σήμερα να τον ευχαριστήσουμε για τη δουλειά του, για τις υπηρεσίες του και να του ευχηθούμε το καλύτερο για το μέλλον. Κύριε Γενικέ Γραμματεύ, αγαπητέ Ζήρη, ήρθε στο 2014, φτάσατε το 2014 στην Επιτροπή των Περιφερειών, πριν, λίγο πριν ξεκινήσει η θητεία αυτή που λίγη σύντομα και για μας. Με μεγάλη χαρά λοιπόν συνεργαστήκαμε μαζί σας, τόσο ο πρώτος αντιπρόεδρος Μάκουλα όσο και εγώ ίδια. Τα τελευταία πέντε χρόνια ηγηθήκατε της Διοίκησης της Επιτροπής των Περιφερειών. Μαζί σας μπορέσαμε και να εξυγχρονίσουμε το, τις μεθόδους εργασίας μας, να ανανεώσουμε το, την Επιτροπή των Περιφερειών, να βελτιώσουμε τον αντίκτυπο του έργου μας σε σχέση με τα λοιπά θεσμικά όργανα. Και επίσης ακολουθήσατε μια γραμμή πιστής υπηρεσίας όλη αυτή τη σταδιοδρομία ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή αλλά και μετά στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η προσωπική σας πορεία σηματοδοτείται από ένα βαθύ ρήγμα μεταξύ ε, Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Ένα βίωμα το οποίο εσείς ως παιδί που γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία αλλά μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία μπορέσατε να το ε, μετατρέψετε σε πλούτο και γίνατε ο καλύτερος πρεσβευτής της διασυνοριακής συνεργασίας που άλλωστε θα ε, παρακολουθήσουμε τις οποίες θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές μέρες και πάλι. Και Είμαι βέβαιος ότι με την ίδια προσήλωση θα συνεχίσετε και μετά την αποχώρηση σας από την θέση αυτή, έστω και με διαφορετικό τρόπο. Σα ευχόμαστε καλή υγεία, να μπορέσετε να απολαύσετε τη συνταξιοδότηση, τη σύνταξή σας, τη εξοδότησή σας, να μπορέσετε να αφοσιωθείτε σε νέα σχέδια και σας παρακαλώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου να δεχθείτε ένα δώρο μικρό, όχι σπουδαίο, βαρύ όμως και βαρύνων. Ένα βιβλίο που περιγράφει, την, ε, περιγράφει με μία φωτογραφική έκθεση την, ε, τις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Euh, αγαπητέ Γύρι, πριν σας ε, δώσω το λόγο, ε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και σας εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι διαλέξετε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Καρλ Χάιντς, αγαπητοί κυρίες και κύριοι μέλη και συνάδελφοι της Επιτροπής των Περιφερειών, με συγκινούν πολύ τα λόγια σας και με ενθαρρύνουν Χαρά και τιμή ήταν η συνεργασία μαζί σας και όπως είπατε κι εσείς αποτέλεσε και μια καμπή στην προσωπική μου ζωή αλλά και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία ο συνδυασμός των βιωμάτων μου και μπορώ να πω ότι ξεκινώντας εδώ και με την ε, εναρκτήρια ομιλία όταν αναλάμβανα καθήκοντα διατύπωσα την παρατήρηση ότι όσοι έχουν εργαστεί σε διασυνοριακό επίπεδο αλλά όπως και σε μένα στο τριεθνές μεταξύ Τσεχίας, Γερμανίας και Αυστρίας έχουν μια διαφορετική σκοπιά, μια σκοπιά που τους επιτρέπει να ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία και έτσι βέβαια δεν μπορώ και, να, και παρά να ε, συνεχίσω στο μέλλον πέραν των καθηκόντων που κατέχω τώρα πάνω στην ίδια γραμμή. Επιτρέψτε μου δύο-τρεις παρατηρήσεις και συνεχίζω στα αγγλικά. Με τρεις παρατηρήσεις λοιπόν που χρειάζεται πιστεύω να τονίσουμε από κοινού και χάρη και στη δική σας την καθοδήγηση κύριε Πρόεδρε και την ε, καθοδήγηση των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, των μελών κτλ έχουμε νομίζω να τονίσουμε πως ε, ήταν και είναι κύρια, ε, κύριο έργο μας η υποστήριξη του δικού σας έργου, των δικών σας θέσεων. Εσείς είστε εκείνοι που ε, έχετε εκλεγεί και περιβληθεί την εμπιστοσύνη του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και άρα καθήκον μας ήταν να σας υποστηρίξουμε και με δύο δρόμους και σε συνεργασία με τους συναδέλφους ε, του θεσμικού οργάνου προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε φέρει πίν με το One Stop Shop που στόχο έχει να σας εξυπηρετήσει καλύτερα να σας διευκολύνει το έργο ένα καλύτερο σύστημα επικοινωνίας μαζί σας μπορέσαμε να ε, θεσπίσουμε αλλά ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να δώσουμε πιο πολύ ουσία στην ε, ε, επικοινωνία με εσά, στην ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας και τη συνεργασία. Θα το είδατε φαντάζομαι πριν από τέσσερα χρόνια όταν κάναμε τις μεγάλες αλλαγές με την υποστήριξη επίπεδο εμπειρογνωμόνων η οποία πήρε πολύ μεγαλύτερη έμφαση διπλασιάστηκε ουσιαστικά η βάση των εμπειρογνωμόνων και έχουμε ακόμα και ένα άλλο στοιχείο. Είναι σημαντικό να σας, ε, το ότι μπορούμε να σας υποστηρίξουμε εξηγώντα και το μοναδικό δυναμικό που έχετε να προσφέρετε ως το ρητή ε, τοπικά εκλεγμένη σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Η επικοινωνία λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έχετε παρακολουθεί στη διαδικασία αυτή ε, όπου προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε δεσμούς και συνεργασίες ε, σε όλη την Ευρώπη οι οποίοι στόχο είχαν να σας επιτρέψουν να αναπτύξετε το δυναμικό σας, το δυναμικό αυτής της εμπιστοσύνης με την οποία έχετε περιβληθεί και να το μεταδώσετε και στα λοιπά θεσμικά όργανα και με αυτό να σταθείτε δίπλα τους. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά. Ε, πάντα στο μυαλό μας το δυναμικό της διοργανικής επικοινωνίας και της βελτίωσης και της ενίσχυση των εργαλείων επικοινωνίας που δεν θα περιορίζονται μόνο στι ευρωεκλογέ. Ένα άλλο σημείο, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς κύριε Πρόεδρε, αλλά και όλους τις κυρίες και κυρίους ε, μέλη κεφαλής των πολιτικών ομάδων κτλ. Γιατί είχα την ευκαιρία εδώ να συναντήσω ένα επίπεδο προσήλωσης αφοσίωσης. Ξέρω ότι πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν χρειάζονταν καθόλου σπρόξιμο για να δουλέψουν. Έχω δουλέψει και σε επίπεδο επιτροπή, έχω εργαστεί και σε επίπεδο εθνικό, αλλά και στο Συμβούλιο σε θέματα αντίστοιχα και μπορώ να πω ότι μπορώ να συγκρίνω. Υπάρχουν λοιπόν παντού άνθρωποι με πολλά κίνητρα και αφοσίωση στη δουλειά του, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με πολύ υψηλό επίπεδο αφοσίωση και προσήλωση και αυτό νομίζω μπορούμε να το αναγνωρίσουμε και στο γεγονό ότι το ότι, το, ότι αντανακλάται αυτό και στο ερωτηματολόγιο ε, αξιολόγησης της δουλειάς που έκαναν οι ίδιοι, τα ίδια τα μέλη και το οποίο νομίζω καταδεικνύει τη σημαντική αυτή αφοσίωση στο έργο σας και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο και η συνεργασία μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων και του προσωπικού και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προσωπικό για την πολύ αποτελεσματική δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και θα περάσω με μια τρίτη παρατήρηση σε ένα πιο προσωπικό ε, θέμα. Είπατε ότι ίσως είναι τα προσωπικά μου βιώματα αυτά τα οποία με οδήγησαν στην Επιτροπή των Περιφερειών εν τέλει. Από το 68 και μετά την εισβολή δηλαδή στη χώρα μου Τσεχοσλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακία. Επί 10 χρόνια περίπου ζούσα πίσω από το σιδηρού παραπέτασμα, δεκαετία 70, δεκαετία 80. Από το 68 μέχρι το 89 ήταν πολύ μακρύς ο δρόμος. Και όπως ε, άρχισα με τις παρατηρήσεις μου στην αρχή επισήμανα πως η τοπική ε, ήταν εκείνοι οι οποίοι παρά το σιδηρό παραπέτασμα μπόρεσαν να εξασφαλίσουν πολύ σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές επί παραδείγματι μεταξύ Τσεχοσλοβακίας και ε, Βαβαρίας πανεπιστήμια και διασυνοριακές συνεργασίες, συνεργασίες. Πράγμα το οποίο με εντυπωσίασε. Ξέρω κύριε Πρόεδρε ότι κι εσείς την ίδια δουλειά προσπαθείτε να κάνετε και σε διαφορετικά επίπεδα Πράγμα το οποίο μου δίνει φτεράκια για το μέλλον. Δύο μηνύματα είναι σημαντικά για μένα, με δύο μηνύματα φεύγω από τη θέση αυτή. Η Επιτροπή των Περιφερειών καταρχάς είναι πιο απαραίτητη από ό,τι ποτέ, πιο απαραίτητη από ό,τι ποτέ στο ρόλο του γεφυροποιού γιατί από μια ελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση που γνωρίζαμε είδαμε να συγκεντρώνονται σκοτεινά σύννεφα. Τα γνωρίζετε όλοι. Το Brexit, τα προβλήματα στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, ε, των πιο πλούσιων και των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, προβλήματα σε σχέση με τις δημοκρατικές αξίες της κοινωνίας μας. Και θεωρώ πως θα κληθείτε εσείς και μάλιστα περισσότερο από ό,τι ποτέ και σε αυτό επικαλούμε και τον Αντιπρόεδρο Έτιγκερ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίο σε πρόσφατη συζήτηση με εμά είπε: Πρέπει, συνάδελφοι, να προετοιμαστείτε για τον αγώνα προάσπιση των δημοκρατικών αξιών περισσότερο από ό,τι ποτέ, σχεδόν με ε, ζώνε ασφαλεία. Και στον ζώντα βλέπουμε τα σύννεφα να πυκνώνουν. Έτσι λοιπόν, και με δεδομένα σε αυτές τις εξελίξεις, πιστεύω η Επιτροπή των Περιφερειών θα είναι φάρος της αλληλεγγύης των δημοκρατικών αξιών θα είναι πιο πολύτιμη από ό,τι ποτέ η προσφορά της. Φεύγω λοιπόν, αποχωρώ από τις Βρυξέλλες, από την ε, θέση αυτή. Σας διαβεβαιώ όμως ότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω να συνεργάζομαι μαζί σας κατά τρόπο ουσιώδη, ζωτικό στα θέματα αυτά, στις αξίες αυτές. Είναι όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, εγγεγραμμένα στο DNA μου. Και το πνεύμα αυτό το οποίο ε, με χαρά μπόρεσα να ε, ζήσω εδώ σε αυτή την επιτροπή θα το μεταλαμπαδεύσω και στην πατρίδα μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητέ μου γύρι για το μήνυμά σας που μέσω ακριβώς των προσωπικών σας βιωμάτων έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για το μέλλον. Θα μας βοηθήσει οπωσδήποτε να καθορίσουμε τις δραστηριότητές μας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ εκ νέου και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τις προσωπικές σας επιδιώξεις στο μέλλον. Και τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση για τις ε, επιπτώσεις των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής μας. Ε, τονίζω ότι η εργασία μας ε, σε όλες τις επιτροπές μας ήταν υψηλού επίπεδου. Με την ενεργό στήριξη της διοίκησής μας και των πολιτικών ομάδων καταφέραμε να κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο τον στρατηγικό μας σχεδιασμό για να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα και για να μπορούμε να διαπιστώσουμε όλο και πιο ορατή επίπτωση της δουλειάς μας στα πλαίσια του στρατηγικού θεματολογίου της Ένωσης. Το έγγραφο που λάβατε όλοι παρουσιάζει ακριβώ τις λεπτομέρειες. Και παρακαλώ, ποιο θα ήθελε το λόγο επ' αυτού. Ήδη έχω δύο εγγεγραμμένου. οπότε πρώτα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Νικόλα Ντρομποσλάβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή Περιφερειών συζήτησε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της περίοδου 21-27 και εγκρίναμε μια γνωμοδότηση με ευρεία πλειοψηφία στα τέλη του περασμένου έτους όπου στηρίζουμε την πολιτική συνοχή της Ένωσης και αντιτιθέμεθα σε οποιαδήποτε περικοπή των δαπανών για τη συνοχή. Και για την κοινή πολιτική, δεν θέλουμε περικοπές για την ανάπτυξη της υπαίθρου, είμαστε επίσης κατά περικοπών των περικοπών των ε, κοινωνικών ταμείων. Θέλουμε περισσότερη χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παράλληλα ενέκρινε την έκθεσή του για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το ερχόμενο, και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι εντελώς ε, παράλληλα τα πορίσματά τους ε, με τα δικά μας. Πρόσφατα οργανώσαμε ένα ειδικό σεμινάριο στο Ντούμπροβνικ της Επιτροπής μας Κοτέρ για το ίδιο αυτό θέμα, το οποίο σεμινάριο συνδυάστηκε με μια συνδιάσκεψη υψηλού επίπεδου των φίλων της συνοχής που οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κροατικής Δημοκρατίας. Σήμερα εναπόκειται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συνεχίσουν την εξέταση του θέματος αυτού. Δυστυχώς ε, η περαιτέρω επιρροή μας είναι περιορισμένη, αλλά μπορούμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η συνοχή είναι θεμελιώδης πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να παραμείνει. Πρέπει να έχει ε, την ίδια δημοσιοφική κάλυψη μέχρι τώρα, που έχει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και τώρα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο λόγια ε, από πλευρά του συγητού Ράισπερμαν, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι καλό που έχουμε αυτή τη συζήτηση για την επίπτωση των ορμοδοτήσεών μας. Λόγω των συνεχιζομένων διαπραγματεύσεων για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Η έκθεσή μας καταδεικνύει ότι οι γνωμοδοτήσεις μας έχουν ε, πολλή επίπτωση στις θέσεις του Κοινοβουλίου για το Ταμείο Συνοχής. Γιατί η πολιτική μας ε, συνοχής τώρα υπάρχει για όλες τις περιφέρειες. Υπάρχει ισχυρή περιφερειακή διάσταση στο Περιφερειακό Ταμείο. Και έχουμε και ισχυρότερη πολιτική για το διάσταση για το κλίμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να Εφησυχάζουμε. Υπάρχουν πολλά θέματα ακόμη που πρέπει να μα απασχολήσουν. Για παράδειγμα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να καταγγείλουμε την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου για μείωση στο 25%. Οπότε, έχουμε αρκετά θέματα για την Επιτροπή Περιφερειών μας για να κάνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένες ε, προτάσεις και να συνεχίσουμε έτσι την σωστή δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο λόγος Χριστόφ Κλέγζο, στον συνάδελφο Χριστόφ Κλέγζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως ε, θα συνεχίσω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ε, ε, για την επίπτωση που θα έχει, έχουν οι γνωμοδοτήσεις μας στους επόμενους μήνες. Γιατί όπω σα είπα δεν ε, σταμάτησε η δουλειά μα. Δεν έχουν ακόμη ψηφιστεί τα κείμενα από το Κοινοβούλιο και οι λεπτομέρειε εφαρμογή των βασικών κειμένων για την κοινοβουλευτική θητεία που αρχίζει τώρα για παράδειγμα τα δημοσιονομικά και η πολιτική συνοχή, όλα αυτά ακόμη δεν έχουν αποφασιστεί. <clears throat> Θεωρώ λοιπόν <clears throat> ότι η πιο σημαντική εργασία μα είναι ακόμη να γίνει. Έχουμε δυνατότητα να επηρεάσουμε την ολοκλήρωση και εφαρμογή των κειμένων αυτών. Θα ήταν πολύ σωστό λοιπόν εμεί ω Επιτροπή Περιφερειών ή νομοθετικοί εισηγητέ για τα βασικά κονδύλια του προπολογισμού να μπορούσαν να συνεχίσουν ε, ω μόνιμοι εισηγητέ για ένα χρόνο ακόμη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να κερδίσουμε τη μάχη να επηρεάσουμε τις επικείμενες αποφάσεις για το πρόγραμμα εργασιών του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή και τα μέτρα εφαρμογή των διαφόρων αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλους. Ευχαριστώ όσους παρενέβησαν. Νομίζω ότι τεκμηριώσαμε πολύ σωστά την εργασία μας και είναι ελπιδοφόρο το μήνυμα. Δεν πάνε μόνο στα σκουπίδια οι γνωμοδοτήσεις μας. Επηρεάζουν τις αποφάσεις, αλλά πολλά ακόμα μπορούμε να κάνουμε και τονίζω ότι πρέπει να ε, παρακολουθούμε τη συνέχεια που δίδεται στις νομοδοτήσεις μας. Επ' αυτών μπορούμε να εμβαθύνουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση έτσι περαιτέρω. Όπως όλοι ε, έχουμε καμιά φορά την ψευδέστηση ότι το βασικό είναι να ληφθεί κάποια απόφαση η προπαρασκευή της λήψης των αποφάσεων αλλά η ουσία είναι μετά στην εφαρμογή των αποφάσεων και πρέπει να διαπιστώσουμε πώς εφαρμόζονται οι γνωμοδοτήσεις μας. Πρέπει λοιπόν να μελετήσουμε το κείμενο αυτό γιατί είναι ένας καλός οδηγός για το μέλλον. Λοιπόν τώρα να δούμε τη γνωμοδότηση για τη συνοριακή διάσταση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Ο εισηγητής μας είναι ο Ρομπέρτο Τσαμπέτη. Έχετε το λόγο, κύριε εισηγητή. Καλημέρα σε όλους. Οι φυσικές καταστροφές δεν γνωρίζουν ε, σύνορα και άρα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των όμορων περιφερειών για να υπάρχει καλύτερος καταμερισμός των δραστηριοτήτων και του συντονισμού αλλά και της ανταπόκρισης στις έκτακτες ε, συνθήκες με μεγαλύτερη προσοχή στην ε, πρόληψη αλλά και τον περιορισμό των συνεπειών του κινδύνου και εδώ θα πρέπει να έχουμε και σενάρια κινδύνου σε διαπεριφερειακό επίπεδο και κλίμακα ε, πέραν των σύνορων δηλαδή για να προλαβαίνουμε αλλά και για να περιορίζουμε και να βελτιώνουμε την ανταπόκριση σε πιθανές ε, φυσικές καταστροφές. Θα πρέπει επίσης να ε, καταρριφθούν τα εμπόδια στη συνεργασία που μπορεί να προκύπτουν από κανονισμούς και ε, από άλλα προβλήματα ε, και έτσι να υπάρχουν οι πρωτοβουλίες εκείνες και οι νομοθετικές οι οποίες επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών. Στα διαπεριφερειακά έργα θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο ουσιαστική συνεργασία και καθώς η νομοθεσία από το ένα κράτος στο άλλο ε, μπορεί να είναι διαφορετική περιπλέκεται η δραστηριότητα συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών ή εκείνων, εν πάση περιπτώσει, που καλούνται να αναλάβουν δράση την ώρα της κρίσης και του κινδύνου. Ε, μας έχουν ζητήσει τα ενωμένα να εισαγάγουμε στην έκθεση αυτή και μια αναφορά στην εκστρατεία ακριβώς των Ηνωμένων Εθνών που στόχο έχει να καταστήσει πιο ανθεκτικές αυτούς τους κινδύνους, πιο ασφαλείς ε, τις πόλεις, πιο έτοιμες να ε, αντιμετωπίσουν φυσικές καταστροφές και πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε ε, να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι κατά τρόπο ουσιαστικό, να αξιολογούνται από κοινού και να καθίστανται οι κίνδυνοι ε, ορατοί μέσα από μια προστασία που μπορεί να παρακολουθεί και ενδεχόμενα γεγονότα που ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί. Καλύτερος ορισμός λοιπόν των στοιχείων του κινδύνου, η ανάπτυξη δικτύων, δεξιοτήτων, γνώσεων, εξειδίκευσης, διάθεσης ε, δυνατοτήτων αντίδρασης μέσα σε ένα πλαίσιο σχετικά ομοιογενές πέραν των ορίων των περιφερειών είναι απαραίτητο και βεβαίως χρειάζονται βάσει δεδομένων ευρύτατες να είναι γνωστό πέραν των συνόρων των εθνικών τι είδου υλικό υπάρχει, τι είδου εξοπλισμό, τι μπορεί να αξιοποιήσει είτε η πυροσβεστική είτε οι δυνάμει ασφαλεία που αναλαμβάνουν δράση κατά τη διάρκεια τη καταστροφή. Χρειάζεται κατάρτιση, χρειάζεται να υπάρχουν και ε, προγράμματα κατάρτιση και για του νέου, ακόμα και μέσα από τι πανεπιστημιακέ του σπουδέ που να του επιτρέπουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους αλλά και να παράγουν έτσι ανθρώπους ε, ικανούς να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές. Ε, επίσης η αξιοποίηση, η ενίσχυση του σώματος ε, αλληλεγγύης που είναι λίγο γνωστό ε, ακόμα στους νέους μας και, μπορού, και θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο με τρόπο ώστε χάρη στις πρακτικές ασκήσεις να δημιουργηθεί ένα σώμα εθελοντών. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και κατάρτιση του ε, προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των υπευθύνων της τοπικής αυτοδιοίκησης που πολλές φορές δεν γνωρίζουν καν ποιες είναι οι ευθύνε τους και άρα χρειάζεται να ενημερωθούν καλύτερα για να ετοιμάζουν καλύτερα την συνεργασία αυτή και την αντιμετώπιση των των κινδύνων. Πρέπει ε, στις διάφορες περιοχές να υπάρχει καλύτερη συνεργασία για τον εντοπισμό των κινδύνων, να επιταχυνθούν οι, κίνδυνοι, οι χρόνοι αντίδρασης και ε, παροχής βοήθειας να αναπτυχθεί και το λεξιλόγιο η ιδιόλεκτος αυτή και με, τις, ε, και με τα αρκτικόλεκτα αυτά που χρειάζονται για να υπάρχει η ταχεία επικοινωνία και η αναγνώριση του κινδύνου από τη μία και από την άλλη πλευρά ε, η ανάπτυξη ειδικών risk manager αρμόδιων, ε, αρμόδιου προσωπικού, προσωπικού αρμόδιου για την αναγνώριση και τη διαχείριση του κινδύνου. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο προσωπικό της Επιτροπής ΕΝΑΤ που μας βοήθησε στην κατάρτιση της ε, γνωμοδότησης, το προσωπικό από την ομάδα μου, την Κιάρα Γκαρμπίνη που είναι η πυρογνώμονας μου, αλλά ταυτόχρονα θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω ε, και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Τζιέκο e ιδιαίτερος για την εξαιρετική συνεργασία, αλλά και την αρμόδια υπηρεσία των ΗΕ που ανέφερα νωρίτερα και η οποία ε, όπως είπα στόχο έχει να προετοιμάσει τον προγραμματισμό ε, του συντονισμού δραστηριοτήτων ε, σε περίπτωση, φυσικό, σε περίπτωση καταστροφών. Και έχω κάποιες τροπολογίες λάβει για τις ιδιαίτερως απομακρυσμένες περιοχές. Έχω προτείνει κάτι πιο ε, συναφές με το κείμενό μου σαν αντιπρόταση προς τους συντάκτες και επίσης έχουμε και την πρόταση του κυρίου Αρμάου που ξέρω όμως ότι ουσιαστικά ζητά ο κύριος Κατάνεο που προσπαθούμε με μια προφορική τροπολογία να προσαρμόσουμε στο κείμενο το αρχικό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που με συνέδραμαν σε αυτή τη διαδικασία επεξεργασία της ε, γνωμοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει η συζήτηση με πρώτον τον Ζωζεφ Μπερίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί η γνωμοδότηση πραγματικά μιλάει για ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Η περιοχή από την οποία κατάγομαι, η Σλοβακία, είναι κοντά στο Δούναβι. Είναι μεγάλο ποτάμι, αλλά και με άλλα μικρότερα ποτάμια ε, είναι υπεύθυνοι για πλημμύρες στην περιοχή μας. Ε, ενίοτε λοιπόν έχουμε ζήσει ε, τέτοιου είδους φαινόμενα και ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε σωστικά συνεργεία, πυροσβεστική, ιατρικές μονάδες κτλ. Αν ζητήσει βοήθεια η περιφέρειά μας, η κεντρική κυβέρνηση δέχεται το αίτημα αυτό και το στέλνει σε μια άλλη περιοχή, σε μια άλλη κεντρική κυβέρνηση, αλλά αργεί δηλαδή να έρθει η βοήθεια. Θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε αυτές τις καθυστερήσεις. Στηρίζω λοιπόν αυτή τη γνωμοδότηση γιατί ενισχύει ε, την ε, διασυνοριακή συνεργασία σε ε, θέματα πολιτικής προστασίας και σίγουρα θα βοηθήσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περίπτωση τέτοιων εκτακτών καταστάσεων ώστε όχι μόνο η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών να διευκολύνεται ε, ώστε να παρέχεται βοήθεια ιδίως εντός ε, του χώρου Σέγγεν αλλά και οι γιατροί, οι πυροσβέστες να μπορούν πιο εύκολα να φτάνουν ε, στο σημείο που τους χρειάζονται. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει η γνωμοδότηση. Ο κύριος Γιάκομπ έχει τώρα το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της ε, γνωμοδότησης αυτής. Αυτό και λόγω της προσωπικής εμπειρίας μου, καθώς ε, είμαι από την ε, περιοχή της Βενέτσια Τζούλια, η οποία γνώρισε ένα μεγάλο σεισμό ε, μέσα στη νύχτα είδαμε να παραβιάζονται όλες τις διεθνείς συνθήκες από το γερμανικό και αυστριακό στρατό για να έρθουν να προσφέρουν βοήθεια στη διάσωση των σεισμόπληκτων το 1962 και θέλω να επισημάνω ότι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα καλούνται να αναλάβουν δράση σε μια περίπτωση καταστροφής οι τοπικοί ερετή με την οργάνωση της διάσωσης σε μια κατάσταση κρίσης που δεν μπορεί παρά να είναι σε ύψιστο επαγγελματικό επίπεδο και πρέπει να έχει περιγραφεί με πολύ λεπτομερούς ρίσκ κανόνες ώστε ο καθένας να μπορεί να ξέρει από την πρώτη στιγμή τι έχει να κάνει. Υπάρχει αυτή η διάσταση λοιπόν ότι αναλαμβάνει δράση πρώτα η τοπική αρχή Ταυτόχρονα όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υπογράμμισε ο κύριος Τσαμπέτη, στόχο έχει και επιδίωξη να δημιουργήσει, να, ε, να εξασφαλίσει τη δημιουργία περιφερειών που θα είναι ανθεκτικές στις καταστροφές αυτές χωρίς να περιορίζονται σε εθνικά σύνορα καθώς τα φυσικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές ξεπερνούν τα πολιτικά σύνορα των εθνικών κρατών και αναφέρονται, αναπτύσσονται σε μια γεωγραφική περιοχή. Και εδώ η ιδιαίτερη ε, έμφαση έχει δώσει και υποστήριξη η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτη. Ευχαριστώ πολύ κύριο Μπλό. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας και βλέπουμε ότι όταν έχουμε αρμοδιότητα ή ευθύνη σε μια διασυνορική περιφέρεια ε, πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να ε, παράσχουμε βοήθεια σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Πυρκαγιές για παράδειγμα στα Πυρηναία μεταξύ του Λαγκτόκ, ε, Οξυτανίας και Καταλωνίας. Ε, έχω βιώσει τέτοιες πυρκαγιές και πραγματικά ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να υπάρχει συνέργεια, σύμπραξη για την αντιμετώπιση από κοινού τέτοιων φυσικών καταστροφών. Το πρόβλημα λοιπόν που τίθεται σήμερα έχει να κάνει και με το εθελοντικό σώμα πυροσβεστών για παράδειγμα και την ετοιμότητά του. Σε πολλά διαμερίσματα στη Γαλλία, σε πολλούς νομούς στη Γαλλία έχουμε θελοντές πυροσβέστες που ουσιαστικά είναι ε, η πλειονότητα. Ε, σίγουρα πλαισιώνονται από επαγγελματίε, αλλά είναι περισσότεροι από αυτούς. Ε, σήμερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας υπάρχει ένας κίνδυνος. Αυτοί οι εθελοντές πυροσβέστες να πάρουν καθεστώς μισθωτού με αποτέλεσμα να ε, υπάρξει πρόβλημα και αβεβαιότητα ε, σε ό,τι αφορά το επάγγελμα ε, του πυροσβέστη. Στην έκθεσή σας μιλάτε για την κινητοποίηση των νέων στο πλαίσιο αλληλεγγύη. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κείμενα που θα θέτουν σε αυτή τη δυνατότητα κινητοποίησης. Πάντως, θέλω να σας δώσω ένα μεγάλο μπράβο για την έκθεσή σας και νομίζω ότι όλοι μας ε, λαμβάνουμε υπόψη τη σημασία που έχει η δυνατότητα αυτή της κινητοποίησης. Πρόεδρος. Ντονάτο το επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε περιφερειάρχης μιας μικρής περιφέρειας που έχει πληγεί από πολλές φυσικές καταστροφές, σεισμούς, πυρκαγιές που δεν μας αφήνουν και πολύ περιθώριο για να οργανωθούμε και καθώς βρισκόμαστε από την Αδριατική έχουμε ως ε, γειτονικές περιφέρειες περιφέρειες της Βαλκανικής. Άρα λοιπόν ε, έχουμε κάποιους περιορισμούς στις, στη δράση μας, στον τρόπο οργάνωσης των δράσεων μας. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτά να αναφερθώ ευχαριστώντας πρώτα τον ε, εισηγητή κύριο Τσαμπέτη για μια γνωμοδότηση ιδιαίτερα εξαντλητική αναπτύσσει πολλά θέματα ιδιαίτερα τονίζει την ανάγκη τη, ε, της έγκαιρης ε, παρέμβασης αλλά και τη σαφήνεια των κανόνων, να γνωρίζει ο καθένα ακριβώ τι έχει να κάνει. Σε αυτό ιδιαίτερα θα ήθελα να σταθώ. Και επίση, συμμερίζομαι μία προσέγγιση που στόχο έχει να ε, καταρρύψει τα πολιτικά σύνορα μεταξύ των ε, ε, όμορων περιφερειών και θα υποστηρίξω βέβαια την γνωμοδότηση αλλά με σημαντικές επιφυλάξεις αυτή τη φορά πρέπει να το πω Ευχαριστώ πολύ δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο το λόγο, οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μα. E- Ευχαριστώ πολύ. Και πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο με στήριξε στη δουλειά μου και με ενίσχυσε στη δουλειά μου είναι η, το ότι ξεκινώντα αυτή την έρευνα ανακάλυψα πως υπάρχουν ήδη συνεργασίε που λειτουργούν παραδείγματι στα όσα ο κύριο Γιάκομ. Υπάρχει μια πολύ κανή συνεργασία μεταξύ της ε, Τζούλια και της ε, Σλοβενία. και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαδοθεί και να συνεχιστεί. Πολλέ είναι οι περιοχέ που έχουν τέτοια συνεργασία, αλλά πολλέ είναι και οι άλλε περιπτώσει όπου κανεί δεν γνωρίζει, όπου κάποιο δεν γνωρίζει από την άλλη μεριά των συνόρων τι υπάρχει και τι μπορεί να αξιοποιηθεί. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε τη δυνατότητα για συνεργασία. Στο συνάδελφο κύριο Μπλαν, Μπιάνκο, θα ήθελα να πω ότι δεν κάνουμε κανένα συμψηφισμό μεταξύ επαγγελματιών και ε, εθελοντών στον κύριο Μπλον διότι βεβαίως έχει τη δουλειά του ο επαγγελματίας αλλά ταυτόχρονα την ώρα της κρίσης ε, την ώρα που εκδηλώνεται η φυσική καταστροφή έχει τεράστια σημασία η προσφορά του εθελοντή χωρίς τους εθελοντές πολλά πράγματα θα είχαν πάει πολύ πολύ χειρότερα δεν ε, θέλουμε σε, με κανέναν τρόπο να περιορίσουμε ή να παρεμποδίσουμε την εθελοντική προσφορά. Αντιθέτω, θέλουμε να την ενισχύσουμε και μάλιστα θέλουμε και σε ασκήσει κοινέ με ε, γειτονικέ χώρε και αντίστοιχα σώματα που θα μα βοηθούσαν να αντιμετωπίσουμε του ε, κινδύνου να ε, δώσουμε περισσότερη έμφαση. Είπα ότι οι ε, εθελοντέ είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να κάνουν ένα άλλο επάγγελμα, επαγγελματικά να έχουν μια άλλη δραστηριότητα, αλλά να είναι, είναι κρίσιμη η συμβολή του στην ώρα της, ε, του κινδύνου, την ώρα της εκδήλωσης φυσικής καταστροφής. Δεν κάνουμε λοιπόν σύγχυση μεταξύ της έννοιας του επαγγελματία, της ομάδας κρούσης ε, που πάντα υπάρχει όταν χρειάζεται την ώρα του προβλήματος, αλλά και του εθελοντή που επίσης θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κινδύνου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Ξεκινούμε με τροπολογία παρθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του που αντικαθιστά την αρχική τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται τροπολογία 3 του εισηγητή, η οποία αντικαθιστά την αρχική τροπολογία 3 και για την οποία υπάρχει προφορικό συμβιβασμό ε, που βλέπετε στην οθόνη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 του εισηγητού αντικαστά την 5 την αρχική υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές, μάλλον εγκρίνεται. Τροπολογία 8 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ της γνωμοδότησης. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται ομόφωνα εγνωμοδότηση συγχαρητήρια στον εισηγητή για το πολύ καλό αυτό αποτέλεσμα. Και περνάμε στη γνωμοδότηση για έναν ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την πτάχη της ανάπτυξης ε, των ε, ναυτιλιακών βιομηχανιών θα δώσω και τη σκητάλη της Προεδρίας ε, Μάρκου Μάρκουλα διότι πρέπει να υποδεχθώ τον Επίτροπο. Θα τα πούμε σε λίγο. Okay, um, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, να προχωρήσουμε λοιπόν. Είδα τον συγητή μας να είναι ήδη έτοιμος. Ο κύριε Κλερζό, έχετε το λόγο να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησία. Σε ευχαριστώ, από πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, που κατέθεσαν τις τροπολογίες τους εμπλουτίζοντας έτσι την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και τον εμπειρογνώμονα ε, που είναι δίπλα μου και τους άλλους συναδέλφους. Ε, λίγοι μήνες απομένουν από τη συγκρότηση της Νέας Επιτροπής. Θέλουμε ακόμα να μπορέσουμε να πειράσουμε τον οδικό χάρτη. Έχουμε μπροστά μας κάποια ζητήματα σημαντικά, ιδίω το γεγονός ότι απουσιάζει εντελώς το ζήτημα των ναυτιλιακού κλάδου. Η γνωμοδότηση αυτή και ιδίω η συνέχεια που θα τη επιφυλάξει η Κομισιόν είναι μια δοκιμή. Ένα τεστ που θα τεστάρει ε, το πόσο θαλάσσιε βιομηχανίε, ο ναυτιλιακό κλάδος θα είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Θα δοκιμαστεί και η αξιοπιστία τη Κομισιόν ε, σε ό,τι αφορά την ανάγκη δημιουργία μια νέα βιομηχανική πολιτική. Αν πράγματι υπάρχει αυτή η βούληση τότε θα πρέπει η ε, ναυτιλιακέ αυτές μηχανίες να έχουν συγκεκριμένο ρόλο λειτουργικό επιχειρησιακό ε, με ορίζοντα το 2030. Η ε, νέα πολιτική στον τομέα τη βιομηχανία το είδαμε ε, και με την έκθεση με έτσι χθε. Ε, δεν περιμένουμε να ακούμε πια. Ε, χρησιμοποιήστε τα εφιστάμενα εργαλεία και αν θέλετε ειδικέ δράσει, ε, αποδείξτε μα ότι τι χρειάζεστε οπωσδήποτε. Γιατί με τέτοιο είδου λογική θα περιμένουμε πάρα πολύ και οι βιομηχανίε θα έχουν στο μεταξύ αφανιστεί. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δούμε ποιε είναι σήμερα οι βιομηχανικέ προκλήσει και να προβλέψουμε ήδη από τώρα προσαρμοσμένα εργαλεία, προσαρμοσμένα ανάστηση στις ιδιαιτερότητες ε, του κλάδου και μιλώ ιδίως για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό θα δοκιμάσει και το πόσο να αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι την ανάγκη να εξελιχθεί η εμπορική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισμού ώστε να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε Ευρωπαίους πρωταθλητές. Τέλος, θα δοκιμάσει και τη δυνατότητά μας και την ικανότητά μας να χρησιμοποιήσουμε τον αυτιλιακό κλάδο για ε, να έχουμε εξυγχρονισμό της πολιτικής σε προστασία του κλίματος, ανακύκλωση πλαστικών, μείωση εκπομπών, οξυδίου, μείωση χρήση του τα κτλ. Με την ευνομοδότηση αυτή μιλούμε επίσης για την πρόκληση ε, που συνιστά η προσέλκυση των νέων ανάπτυξη ε, των ακτών, ε, των παράκτων περιοχών και βιώσιμη ε, ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Θέλουμε επίσης βελτίωση των δεξιοτήτων και γι' αυτό θέλουμε να υπάρξουν ευρωπαϊκά δίκτυα, σύντεκο e τα λέμε, για να βοηθηθεί η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και να υπάρξει διαπεριφερειακή συνεργασία. Ίσως εκπλήσονται ορισμένοι ε, από τον αριθμό των τροπολογιών που κατέθεσα εγώ προσωπικά. Χρειαζόταν όμως αυτό, γιατί ήθελα να λάβω υπόψη ε, τις ε, προτάσεις των διαφόρων ενδιαφερομένων. Τέσσερι μήνε πάει που το συζητήσαμε στην Επιτροπή ΝΑΤ. Ε, έκτοτε ε, κατητέθηκαν πολλέ τροπολογίε ε, που ζητούν να επενδύσουμε σε παραδοσιακού παράγοντε ηθαιοκαλλιέργεια και πρέπει και αλίας. Ε, σίγουρα μιλάμε για την γαλάζια οικονομία. Τομεί πάρα πολύ σημαντικοί λοιπόν αυτοί οι δύο και από τώρα πρέπει να επενδύσουμε. Έχουν επίση επιμείνει πολλέ τροπολογίε στην ανάγκη μια ειδική προσέγγιση για τον αφιλιακό την υποστήριξη των λιμένων, ιδίω στις από απόκεντρε περιφέρειες και συμπεριλαμβάνω στου τροπολογισμούς τι πολύ σημαντικέ αυτέ προτάσει. αγαπητοί συνάδελφοι. Περιμένω τι παρατηρήσει σα στην ψηφοφορία με ε, θετική ε, διαδικασία διάθεση και αισιοδοξία. Ελπίζοντας ότι θα ε, ευοδοθεί η προσέγγιση που προτείνουμε με την γνωμοδότησή μας, ε, γιατί είναι μια τομιακή προσέγγιση η οποία ε, τρέχει πολλέ πολιτικέ, αφορά το πεδίο αρμοδιότητα πολλών από τι επιτροπέ μα και θα επηρεάσει σίγουρα το μέλλον των παράλληλων περιοχών σε πολλέ από τι χώρε μα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή αυτή. Υπάρχουν παρεμβάσεις από την αίθουσα. Εσείς εκεί πίσω. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την τροπολογία 16. Θα την καταψηφίσει σου ειδική αντιπροσωπεία απλά και μόνο γιατί όταν γίνεται λόγος για συγκεκριμένες μόνο περιφέρειες ε, ε, αποκλείεται κάποιες άλλες. Αυτό αφορά συναδέλφους από τη Φιλανδία, την Πολωνία, τις χώρες της Βαλτικής. Γιατί η περιοχή της Βαλτικής ε, χρήζει ειδική προσέγγισης. Γι' αυτό ήθελα να σας εξηγήσω ότι ε, παραγνωρίζετε κάτι που είναι σημαντικό, ε, την ιδιαιτερότητα δηλαδή του περιβάλλοντος της Βαλτικής, εξού και εμείς θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ να κατάλαβα καλά. Αναφερθήκατε στην τροπολογία 16, η οποία όμω έχει αποσυρθεί μετά από διαπραγματεύσει των δύο πολιτικών ομάδων. Οπότε δεν χρειάζεται να την καταψηφίσετε. Αυτά που είπατε για τη Σουηδία, Φιλανδία και άλλες χώρες, όλα αυτά ε, τα λάβουμε υπόψη και ε, αποσύρθηκε η τροπολογία. Υπάρχει καμία άλλη παρέμβαση. Αν όχι, τότε να ψηφίσουμε. η τροπολογία 1R του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά δεκτή. Και καταπίπτει η 1. Λοιπόν, μετά ψηφίσουμε μαζί τις 2 ε, και 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά δεκτές. Τροπολογία 4, ο εισηγητής είναι υπέρ είναι δική του πρόταση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτή. Πέντε. Ο ζητητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε από κοινού 6 έως 9. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτές. Τροπολογία 10. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτή. Η τροπολογία του εισηγητή 11R. Υπέρ παρακαλώ. Α, ε, κύριε εισηγητα θέλετε να εξηγήσετε κάτι για την τροπολογία σας, παρακαλώ. Ναι, τονίζω ότι η τροπολογία αυτή ε, παρουσιάζει στην θέση μα, την προσέγγιση μα για το διεθνέ εμπόριο, μετά από τροπολογία Γκαμαλό Αλέ στη Μάλτα, τονίσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί από αθέμητο ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα πρέπει να επιλέγει τι πολυμερεί διαπραγματεύσει για το ελεύθερο εμπόριο εκεί που είναι αποτελεσματικέ. Και βεβαίω οι Έλληνε φίλοι είχαν προτείνει μια πολύ ισχυρή φιλελευθερωποίηση των ε, ναυτιλιακών υπηρεσιών που αντιτίθεται στο συμβιβασμό της Μάλτας. Είπα ότι πρέπει να επεκταθεί η τροπολογία και στις ναυτιλιακές υπηρεσίες, όχι μόνο στην ναυτιλία, αλλά ε, να κρατήσουμε το συμβιβασμό που είχαμε επιτύχει στη Μάλτα. Ευχαριστώ για την ε, διευκρίνηση αυτή. Η, τροπολογίες, η τροπολογία αυτή καλύπτει τις τροπολογίες 11 13. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ τις τροπολογίες του εισηγητή. Ευχαριστώ κατά. πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Can we close the vote? Πέρασε. Α, όχι. Ωραία, τώρα πέρασε. Η πλειοψηφία είναι υπέρ, εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 11, 12, 13 καταπίπτουν. Κατόπιν από κοινού 14 και 15. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 16 αποσύρθηκε όπως είπαμε. 17, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτή. 18 υπέρ παρακαλώ. Κατά. 19 άρα. Είναι τροπολογία του συγητή που καλύπτει την τροπολογία 19. Υπέρ παρακαλώ τη τροπολογία του συγητή. Κατά. Δεκτή. Καταπίπτει 19. 20. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 21. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Λοιπόν, 22R του εισηγητή υπέρ παρακαλώ κατά δεκτή 22 r του εισηγητη υπερ παρακαλω κατα δεκτη 22 πιπτη 23 Συγητής είναι κατά Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ Κατά Απορρίπτεται Από κοινού προτείνω από την 24 έως την 31 υπέρ παρακαλώ κατά δεκτές 32 υπέρ παρακαλώ κατά δεκτή 33R του εισηγητή που καλύπτει 33-34. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτή. Οι 33 και 34 καταπίπτουν. 35 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτή. Από κοινού. 36 έως 42 υπέρ παρακαλώ κατά δεκτές η τροπολογία 43R του εισηγητή υπέρ παρακαλώ κατά δεκτή 44. R, Τροπολογία του συγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτή. 44-45 καταπίπτουν. Η τροπολογία του συγητή 46R. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτή. 46 και 47 καταπίπτουν. Ωραία. Τελική ψηφοφορία για την τροποποιηθήσα γνωμοδότηση υπέρ παρακαλώ κατά μία ψήφος κατά αποχές δύο με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίνεται αυτή η γνωμοδότηση και συγχαίρουμε τον εισηγητή μας. Right, let's take the Οπότε, επόμενη γνωμοδότηση. Πολυπίπεδη διακυβέρνηση και διατομιακή συνεργασία για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Καλωσορίζω την κατατότητα. Παρακαλώ, παρουσιάστε την γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία Πολλά λέμε για την ενεργειακή μετάβαση. Αλλά δεν αναφερόμεθα στο ποιο θα πληρώσει το λογαριασμό αυτή τη μετάβαση. Πάνω από 50 εκατομμύρια Ευρωπαίων έχουν δυσχέρειε κάθε χειμώνα να πληρώσουν ε, το λογαριασμό θέρμανση ε, του σπιτιού του. Πάνω από 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν σε ε, σπίτια τα οποία είναι να δεν έχουν μονοθεί, έχουν υγρασία. Οπότε στόχος μου είναι να επιστήσω την προσοχή ημών και ημών για να δείτε τι μπορείτε εσείς ως πόλεις, ως τοπικά εκλεγμένοι, ως δήμαρχοι να κάνετε. Διότι οι κυβερνήσεις μας αργούν να αντιδράσουν για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό της ενεργειακής πτώχειας. Δεν υπάρχει ούτε καν ε, δεσμευτικός ορισμός. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως τοπικά εκλεγμένοι. Πολλά, πολύ περισσότερα. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να ε, εντοπίσουμε τα άτομα αυτά που έχουν αυτό το πρόβλημα. Και δεν ξέρουμε ποια ακριβώ είναι. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι δεν είναι μόνο κοινωνικό αυτό το θέμα. Γιατί αυτό που θα κάνουμε σήμερα για τα προβλήματα των χαμηλών εισοδημάτων, ε, της έλλειψης μόνο στα σπίτια, των υψηλών τιμών της ενέργειας, όλα αυτά δεν είναι μόνο θέματα κοινωνικά. Είναι επίσης περιβαλλοντικό θέμα. Γιατί πολλοί, για παράδειγμα, καίνε απόβλητα εντός ε, του μοναδικού δωματίου του σπιτιού το οποίο προσπαθούν να θερμάνουν. Πρέπει λοιπόν σε τοπικό επίπεδο να έχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση. Γνωρίζω ότι περισσότεροι γνωρίζετε την σύμβαση των δημάρχων. Είναι ένα κίνημα δημάρχων που προσπαθούν να προωθήσουν την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Αυτή η σύμβαση έχει ως τρίτο πυλώνα της δράσης της την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Αν εσείς ως τοπικά εκλεγμένοι θέλετε να ενταχθείτε σε αυτό το δίκτυο, να ανταλλάξετε απόψεις για το θέμα αυτό, να μάθετε από άλλες πόλεις, από την εμπειρία τους, παρακαλώ να ενταχθείτε σε αυτή τη σύμβαση δημάρχων, έτσι θα καταλάβετε ποιο είναι το θέμα, θα βρείτε βέλτιστες πρακτικές, καλές μεθόδους, πώς να εντοπίσετε τα προβλήματα που υπάρχει ενεργειακή φτώχεια και μπορείτε να αξιοποιήσετε και το παρατηρητήριο ενεργειακής φτώχειας και εκείνοι μπορούν να σας στείλουν στοιχεία για να σας βοηθήσουν στη δουλειά σας. Θέλω λοιπόν να αντιληφθείτε ότι είναι καθήκον σας και αυτό. Πρέπει να βοηθήσετε τα άτομα να γίνουν από παραγωγή ενέργειας να βοηθήσετε όλους σας τους συμπολίτε να έχουν σπίτια που να μπορούν και να έχουν θέρμανση και να έχουν ε, κλιματισμό. Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι εμπλέκονται στα ενεργειακά θέματα. Σε ευχαριστώ πολύ για τις τροπολογίες σας. Χαίρετε. Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ που μας υπενθυμίσατε ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Έχουμε καθήκοντα λοιπόν. Λοιπόν, θέλει κανείς τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την κυρία Τούτα για αυτή την γνωμοδότηση. Ο ρόλος μας ως ε, τοπικών και περιφερειακών φορέων είναι να ε, αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Όντως, ε, στη γνωμοδότησή σας αναφέρεται τα τρία βασικά θέματα. Είναι η ενεργειακή φτώχεια, τα χαμηλά εισοδήματα και οι υψηλέ τιμέ ενέργεια. Όλα αυτά μα ενδιαφέρουν. Κυρίω όμω μπορούμε να δράσουμε για την καλύτερη μόνωση των κτισμάτων. Πρέπει όλα τα κτίσματα να γίνουν είτε ενεργειακά παθητικά ή να γίνουν ενεργητικά στην παραγωγή ενέργειας. Μπορούμε να δράσουμε για τα θέματα αυτά. Και γι' αυτό τονίζω ότι αυτά που είπατε πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Ο κύριος Καμπόρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να υπογραμμίσω ένα πρόβλημα που είναι το εξής. Κάθε πλούσιος έχει ένα τζάκι στο σαλόνι και βέβαια είναι ένδειξη πολυτέλεια αυτό. Ο φτωχό όμω με μία σόμπα ή με ένα μικρό τζάκι μπορεί να θερμάνει το σπίτι του μόνο μερικέ φορέ. Και ξέρουμε ότι ε, πολύ συχνά στι φτωχέ περιοχέ ε, τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται είναι κακής ποιότητας στερεά καύσιμα, ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε και ε, πιο συχνά στις, ε, στην Ήπεθρο, στις μικρές πόλεις, όχι στα μεγάλα κέντρα. Έτσι λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε και αυτή τη διάσταση της ενεργειακής φτώχειας. Και ε, περνάω σε ένα άλλο πρόβλημα σχετικό, ότι εάν χρησιμοποιείται ξυλία ως πηγή ενέργειας για τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού δεν θα μείνει αρκετό φθηνό ξύλο καλή ποιότητας για τους φτωχούς, για τα σπίτια τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκαριάννης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια πολύ καλή γνωμοδότηση από τη συνάδελφο. Πρέπει να πούμε ότι Σήμερα μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια λόγω και των κοινωνικών ανισοτήτων. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στι κοινωνικέ ανισότητε γιατί υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί ανθρώποι. Οι πλούσιοι μολύνουν το περιβάλλον με τον πολυτελή και υπερβολικό τρόπο ζωή όπω ζουν σε μεγάλα σπίτια, ε, έχουν μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα, έχουν και θερμενόμενε πισίνε. Ενώ οι φτωχοί κύριε πρόεδρε προσπαθούμε με τρόπους να θερμάνουν τα σπίτια τους με τη χρήση κακής ποιότητας ξύλου για καύση. όλοι μας μολύνουμε το περιβάλλον και ο καθένας με τον δικό του τρόπο και πρέπει να δώσουμε επιτέλους έμφαση στα παιδιά αλλά και στους ίδιους τους γονείς για προστασία του περιβάλλοντος και η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να γίνει επίσης μέρος της καθημερινότητας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ουδή. Εγκρίνεται. Ο συγητή τώρα έχει καταθέσει τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 2. Η αρχική 3, 4, 5, 6 και 7 από κοινού. Ψήφι υπέρ κατά ουδής άρα εγκρίνονται όλες αυτές οι τροπολογίες τροπολογία 8 αρτήσιγη του ψήφι πέρ κατά μία ψήφος κατά εγκρίνεται επομένω. τροπολογία 9 ψήφι πέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 10 ψήφι πέρ κατά Δις εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ψήφι περ. Κατά. Ουδής εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία του συνόλου γνωμοδότης όπως τροποποιήθηκε. Ψήφι περ. Κατά. Ουδής. Αποχές. Ουδία, ουδεμία. Εγκρίνεται ομόφωνα η γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Okay, uh, Commissioner and... Ο Επιτρόπος Κανιέτε και ο Κάρλ Χάιντς Λάμπερτς είναι καθοδόν, οπότε διακόπτουμε για πολύ λίγο. Και θα παραδώσω πάλι την Προεδρία στον Καρλ Χάινς.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

Chers collègues, nous reprenons maintenant la séance. Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναρχόμεθα. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, καταρχάς σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρουσία σας. Εκ νέου, χαίρομαι που συνεργαστήκαμε σε τέτοιο μεγάλο βαθμό την τελευταία πενταετία. Σε ευχαριστώ για τη μεγάλη διάθεσή σας να έρχεστε στην Επιτροπή μας. Επανειλημμένα. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων για την κλιματική, πολιτική, για την περιβαλλοντική και την ενεργειακή της Ένωσης. Είναι μεγάλη χαρά λοιπόν που ε, σήμερα. Πρώτα απ' όλα για να κάνουμε ένα απολογισμό για αυτά τα τόσο έντονα τελευταία πέντε χρόνια και για να δούμε και πώς διαμορφώνεται το μέλλον που θα είναι η βάση της εργασίας ε, του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τη νέα Επιτροπή των Περιφερειών. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία αξιολόγηση τα εθνικά ενεργειακά και κλιματικά προγράμματα, των εθνικών ενεργειακών και κλιματικών προγραμμάτων και ζήτησε σαφώ από τα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερε φιλοδοξίε. Α μην κρυβόμαστε. Πολλά ακόμη πρέπει να κάνουμε. Πολλοί δρόμο είναι ακόμη μπροστά μα για να επιτύχουμε του στόχου μα για το 2030, να οικοδομήσουμε δηλαδή την ευρωπαϊκή στρατηγική για να επιτύχουμε το μακροπρόθεσμο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Ε, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε αποτελεσματικά μόνο εάν ε, κάνουμε ένα διάλογο με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τους συμπολίτε και τους άλλους εμπλεκομένους φορείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να εφαρμόσει τη Συμφωνία των Παρισίων και θα κάνει κάθε προσπάθεια να επιτύχει τους στόχους της η προκαταρκτική διαπραγμάτευση πριν από την επόμενη κόπ που θα ολοκληρωθεί ε, σύντομα στη Βόνη και έχουμε μερικούς μήνες για να προετοιμαστούμε για την COP25. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και των δεσμεύσεών της, αλλά πρέπει να διατηρήσει και την πρωτοπορία της για τα κλιματικά θέματα με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να επιτύχουμε την ε, κλιματική ουδετερότητα, την οποία ε, θέλω να πω ότι η Επιτροπή μα στηρίζει εδώ και πολύ καιρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι η ακμή του δόρατο αυτή τη φιλοδοξία και κύριε Επίτροπε, εκτιμούμε ιδιαίτερα τον πρώτο ρόλο που παίζετε εσεί στον τομέα αυτό. Οι πόλει, οι περιφέρειε, τα χωριά μα καθημερινά μάχονται κατά των επιπτώσεων τη κλιματική αλλαγή. Η δέσμευσή του αξιοποιήθηκε και συντάχθηκε αποτελεσματικά χάρη για παράδειγμα στην επιτυχία τη σύμβαση των δημάρχων. Είναι μια πρωτοβουλία, μια επιτυχία που πρέπει να επιβεβαιωθεί και να διευρυνθεί εν ώψη του ορίζοντο 2030. Οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ είναι στην πρώτη γραμμή για να δώσουν μια πρώτη απάντηση στι αυξανόμενε απαιτήσει των συμπολιτών μα και των επιχειρήσεων για μια πιο βιώσιμη Ευρώπη. Οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ τη Ένωση έχουν ανάγκη από ένα νομοθετικό πλαίσιο φιλόδοξο που να λαμβάνει υπόψη τι εμπειρίε του, τις καλές τους πρακτικές αλλά και τα εμπόδια και τις ανάγκες τους και ε, τις ε, συγκεκριμένες αδυναμίες τους. Χρειάζονται ένα διαμονωσικό πλαίσιο, επαρκή χρηματοδότηση για να τοποκριθούν στις προκλήσεις του κλίματος. Με πολύ χαρά λοιπόν θα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα μαζί σας. Οπότε χωρίς περαιτέρω χρόνο τριβή σας παραχωρώ το λόγο. Αγαπητέ πρόεδρε Λάμπερτ, αγαπητοί συγητέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά που με απευθύνατε σήμερα την πρόσκληση αυτή, αλλά και για την συνεχή επικοδομητική δράση σα για τα θέματα του κλίματο. Πλησιάζει το τέλο τη θητεία τη Κομισιόν και είναι μια κρίσιμη χρονική στιγμή, γιατί πρέπει να αναλυφθεί αποφασιστική δράση για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Πρέπει και να μειώσουμε τι διαστάσει του φαινομένου, αλλά και να περιορίσουμε τι επιζήμιε συνέπειε του. Οι Ευρωπαίοι πολίτε στην πριτρικτική του πλειοψηφία αναγνωρίζουν αυτή την πρόκληση. Είδαμε πρόσφατε διαμαρτυρίε για το κλίμα που δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη ανάληψη δράση. Η ε, κοινή γνώμη μα υποστηρίζει και δείχνει ότι οι πολίτε θέλουν και αυτοί να συνεισφέρουν. Το έργο τη επιτροπή των Περιφερειών είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο. Οι περιφερειακοί τοπικοί φορείς είναι σημαντικοί για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της καθημερινότητας των δράσεων στο επίπεδο ε, του απλού πολίτη. Θέλω να συγχαρώ τους περιφερειακούς και τοπικούς ηγέτες για τη σημαντική δουλειά τους ό,τι αφορά το κλίμα, την ενέργεια, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια έλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες ε, και έτσι οι ηγέτες αυτοί ενώνονται γύρω από ένα κοινό όραμα. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ε, είναι σημαντική για τη δράση ό,τι αφορά το κλίμα. Θα συνεχίσω λοιπόν οι πόλεις ε, και οι Δήμοι να στηρίζουν την επιτεύξη των στόχων ε, του 2030 καθώς και τη Στρατηγική Ένωση για την προσαρμογή της στην αλλαγή του κλίματος. Ε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία, λέγαμε αυτό το σύμφωνο των δημάρχων, εθνικά υπουργεία, περιβαλλοντικοί φορείς κτλ. Πάνω από 9.000 πόλεις έχουν βάλει ποσοτικού στόχου για τη μείωση του επίπεδου διοξιδιωτών θα ξεπάνω από 1.500 πόλεις όπως και ε, στην ανάγκη να υπάρξει να δράσεις προσαρμοστικές. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να ενθαρρύνετε και άλλες πόλεις και άλλους δήμους και περιφέρειες ε, να ενταχθούν σε αυτό το σύμφωνο των δημάρχων. Δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ε, α, ότι θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρεκόρ επιδόσεων. Ε, είμαστε καινοτόμοι, ενθουσιώδεις ε, φορείς. Ε, είναι η στόχη του 2030. Εμείς ε, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ε, βέβαια πάντοτε πρέπει να γίνονται σεβαστοί και οι κανόνες της ιστορικής αγοράς. Το CBU το Μάιο πόλεις από 21 χώρες και από 7 γειτονικέ χώρες απίθανα έκλεισε ο Ευρώπης να είναι φιλόδοξη είναι πολύ σημαντική ε, η ανάληψη κλιματικής δράσης οι πόλεις που είναι και κόμβοι καινοτομία ε, μπορούν να προσφέρουν ε, άμεσες ε, αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις. Επίσης έχουν πολλούς ανθρώπους και πολλά άλλα θετικά ατού αλλά και κινδύνους ταυτόχρονα. Υπάρχει το πρόβλημα της κλιματικής και της κοινωνικο-οικονομικής ευαλωτότητας που αλληλεπικαλύπτονται. Θα πρέπει λοιπόν να χαρτογραφήσουμε τους κινδύνους και ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι είναι σημαντικός αν θέλουμε να υπάρχει αντοχή για τους ευάλωτους πληθυσμούς. Έχουμε ξεκινήσει και κάποιες πρωτοβουλίες, για παράδειγμα για την ενεργειακή φτώχεια, για τις μεταβατικές περιφέρειες που εξορίσσονται ορυκτά καύσιμα, για τις νησιωτικές περιοχές ε, ε, ώστε να χρησιμοποιούν καθαρή ενέργεια. Αντιλάσσουμε εμπειρίε ε, και βέλτιστες πρακτικές. Μπορούμε να βελτιωθούμε γιατί έτσι θα προσφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και δεν θα αφήσουμε πίσω καμιά περιφέρεια. Ταυτόχρονα η κλιματική δράση δεν συμβαίνει μόνο στις μεγάλες πόλεις. Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής είναι προφανής σε όλες τις περιφέρειες, είτε είναι αστικές είτε όχι. Και οι τοπικές κοινότητες την Ευρώπη πρέπει να είναι μέρο τη λύση. Θέλουμε να πετύχουμε μηδενικές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων. Το έχουμε θέσει ως στόχο για το 2050 στην Ευρώπη. Αυτό απαιτεί άμεση δράση όμως εντό και εγκάρσια ε, διάφορου τομεί, σε όλα τα επίπεδα. Θέλουμε μετάβαση γρήγορη, ε, εκτεταμένη στα συστήματα. Ενέργεια, βιομηχανία, χρήση γη, οικοσυστήματα, σχεδιασμός, υποδομέ, Βέβαια και ε, ευρύτερο πλαίσιο που έχουμε εδώ να λάβουμε υπόψη είναι η βιώσιμη στόχη ανάπτυξη. Βέβαια δεν μιλάμε μόνο για ανταπόκριση στις προκλήσεις αλλά και για την ε, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ευκαιριών που θα βοηθήσουν ε, τους πολίτες ε, μέσω της χρήσης νέων θέσεων πιο καθαρού. Αναγνωρίζεται επίσης στη Συμφωνία των Παρισίων ο ρόλος των τοπικών φορέων για την δημιουργία συνεργασίας και ανθεκτικότητας. Θέλω να επαναλάβω λοιπόν τις δράσεις οι οποίες αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μειώσουμε τις θερμοκηπιακές εκπομπές ε, αερίων, για βιώσιμη ενέργεια σε προσιτές τιμές. Είμαστε η πρώτη μείζων οικονομία που έχει ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για να κάνουμε πράξη αλλά και να ξεπεράσουμε τις δεσμεύσεις των Παρισίων. Έχουμε φιλόδοξο στόχο για το 2030 για μείωση αερίων, θερμοκηπίου, ανανόσιμη ενέργεια, ε, ενεργειακή απόδοση, δημιουργία ενεργειακής ένωσης. Έχουμε ένα μοναδικό σύστημα για την κλιματική ε, ενεργειακή διακυβέρνηση ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να μπορούν από κοινού να ε, κάνουν τον προγραμματισμό τους ώστε να πετύχουν τους στόχους του 2030 καθοδόν προς τη μετάβαση σε μια κλιματική πραγματικά ουδέτερη οικονομία που θα είναι δίκαιη για όλους. Θέλουμε επίση και συνοχή για προβλεψιμότητα για τους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας τα κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετήσουν ολοκληρωμένα ε, προγράμματα για την περίοδο από το 2021 στο 2030 για να δείξουν ότι μπορούν να ε, υλοποιήσουν αυτού του στόχου του 2030. Όλα τα κράτη-μέλη υπέβαλαν τα πρώτα τέτοια σχέδια ε, την, πρόσφατα και την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν παρουσίασε τις δικές της προτάσεις και τεχνικές συστάσεις είναι θετικό για την επιτεξία του 2030. Ωστόσο, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο και περιθώρια βελτίωσης, όπως φαίνεται και στις συστάσεις αυτές για τις οποίες σας μίλησα. Πού βρισκόμαστε τώρα λοιπόν. Τα καλά νέα είναι ότι συνολικά η μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου στην Ένωση το 2030 ήδη υπολογίζεται ότι ευθυγραμμίζεται με το στόχο του μείον 40 σε σύγκριση με το 1990. Ωστόσο, δεν έχουμε πετύχει του στόχου μας για το μισό εκτός του σύστημα εμπορία εκπομπών που είναι 28% το 2030 σε σχέση με το 2005 ενώ έπρεπε να είναι 30, μείον 30 δηλαδή της 100. Βλέπουμε επίση μια διαφορά σε ό,τι αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας για τι ανανεώσιμες πηγέ ενέργειας 32 ε, τουλάχιστον ανανεώσιμε σε ό,τι αφορά τελική κατανάλωση ενέργεια και στόχος ε, αποδοτικότητα 32,5. Ε, το κενό σε Τώρα τι ανανεώσιμε έχουμε ε, μικρό ποσοστό γύρω στο 1,6% αλλά για την ενεργειακή απόδοση μεγάλο κενό 6 ποσοστίων μονάδων. Άρα πρέπει να κάνουν παραπάνω προσπάθειε στα κράτη-μέλη. Καλή είδηση είναι ότι έχουν 6 μήνε τώρα για να αυξήσουν το επίπεδο φιλοδοξία στα κράτη-μέλη. Έγινε πολύ σημαντική δουλειά ανάλυση συστάσεων από πλευρά Κομισιών. Έτσι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα κρατη να ολοκληρώσουν μέχρι το τέλο του έτου ε, τα σχέδιά του. Αυτή τη διαδικασία πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχει ε, και ε, το ευρύ κοινό τις δυνατότητες να συμμετέχει για την προετοιμασία των τελικών σχεδίων. Πρέπει να υπάρξουν αλληλεπιδράσεις ε, και να δοθούν απτά παραδείγματα project που θα υιοθετηθούν την επόμενη δεκαετία. Εκ παραλλήλου θα συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε την συμμετοχή όλων των παραγόντων της κοινωνίας με συστημικό τρόπο και θα ενισχύουμε τις συνέργειες σε εθνικό, ευρωπαϊκό, τοπικό επίπεδο. Πέραν του 2030 τώρα. Πέρυσι τον Νοέμβριο παρουσιάσαμε ένα στρατηγικό σχέδιο για μια ουδέτερη οικονομία από κλιματικής πλευράς. Είναι ο δικός χάρτης για την πολιτική της Ένωσης. Αυτή είναι η μακροπρόθεσμη συνεισφορά της Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της ε, Συμφωνίας των Παρισίων. Είναι μια έκκληση σε όλα τα θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια, τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ε, δήμους, ε, κοινότητες και μεταξύ άλλων νεολαία και άλλους φορείς της κοινωνίας. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε επίση και άλλου διεθνεί εταίρου να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την πρόταση τη Κομισιόν για την θέσπιση μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων για κλιματική ουδετερότητα. Μηδενικέ εκπομπέ δηλαδή αεροθερμοκοκυπίου μέχρι το 2050. 20... Τρία κράτη-μέλη ήδη έχουν ε, δεσμευτεί. Κάποια ζήτησαν περισσότερο χρόνο. Συμφώνησε το Συμβούλιο και θα επανέλθει σε μια επόμενη συνεδρίασή του στο θέμα. Θεωρείται ότι είναι σημαντική η πρόοδος εν ώψη του μεγέθους της πρόκλησης. Για του εξή λόγου. Πρώτο, γιατί είμαστε πολύ κοντά. Σχεδόν φτάνουμε. Και φτάνουμε και με το σωστό τρόπο στο σημείο του τερματισμού. Ήδη από τον Νοέμβριο είχαμε πει πέρυσι ότι θέλουμε ευρεία δημοκρατική συζήτηση που θα ε, εμβαθύνει στα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί επιτάπητος ε, και θα κάνουν τα δέοντα και τα κράτη-μέλη. Και το βλέπουμε να συμβαίνει πράγματι στην Ευρώπη. Χαιρόμαστε που μεγάλη πλειοψηφία κρατών μελών έχει καταλήξει και δεν μας εκπλήσει το ότι χρειάζεται συζήτηση σε κάποια ακόμα κατά τη μέλη που θα έχει μια τέτοια επιλογή. Δεύτερη Δεύτερο λόγο για τον οποίο θεωρούμε ότι είναι θετικό είναι ότι εστιάζει η συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πώ θα το πετύχουμε, πώ θα πετύχουμε το στόχο μα, πώ θα έχουμε αυτή την κλιματική ουδετερότητα ε, και μάλιστα ω περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική επιτυχία. Πρόκειται για μια μεγάλη επενδυτική πρόκληση για την Ευρώπη. Έχουμε τι τεχνολογίε, έχουμε του πόρου. Πώ όμω θα του κινητοποιήσουμε στην απαιτούμενη ταχύτητα και μέγεθο, Πού είναι τα κίνητρα Πρέπει να μείνει λοιπόν στο θεματολόγιο ψηλά η κλιματική ουδετερότητα και θα πρέπει να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτή τη δίκαιη ε, και οικονομικά αποδοτική μετάβαση. Έχουμε ξεκινήσει ε, να προωθούμε ε, τους παράγοντες που θα διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση και έχουμε και τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων τους οποίους θα προσπαθήσουν να εφαρμόζουν σε διεθνέ επίπεδο. Ο στόχο μα τώρα περνάει στην εφαρμογή των στόχων Οι διάφορε χώρε ε, ανέλαβαν δεσμεύσει. και πρέπει να έχουμε μια σφαιρική αισιοδοξία. Αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσει τη Ένωση, συναντώνται στη Βόνη με του διεθνεί εταίρου στα πλαίσια τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και συζητούν τους κανόνες για να γίνουν πραγματικότητα οι στόχοι των Παρισίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι σημείο κλειδί για την ε, κλιματική, το κλιματικό θεματολόγιο. Η σύνοδος των ΗΠΑ που θα γίνει το Σεπτέμβριο και μπορεί να προδώσει μεγαλύτερη όθηση στις ε, επιμέρους φιλοδοξίες αλλά και να επιταχύνει τις εξετάσεις και έτσι χρειάζεται οπωσδήποτε οι πόλεις, οι περιφέρειες, όλες οι τοπικές αρχές να συμβάλλουν και να επιταχύνουν το έργο τους. Έχουμε πολύ, έχετε πολύ σημαντική θέση εσείς. Μπορείτε να λάβετε δράση και στις περιοχές σας αλλά και να δώσετε το καλό παράδειγμα ώστε να καθοδηγήσετε τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποσταρίζει τις ε, ε, περιοχές, τις τοπικές οργανώσεις και δομές με ιδιαίτερα ταμεία τα οποία μπορούν να δώσουν έμφαση στο περιβάλλον. παραδείγμα, το 2014-2020 το, το Περιφερειακό Ταμείο πάνω από 100 εκατομμύρια, το μισό του δηλαδή, είχε επενδυθεί σε πόλεις. Επίση, αναγνωρίζουμε πω πρέπει να επιταχυνθεί αυτή η υποστήριξη και για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για ζωτική σημασία ε, οικονομική υποστήριξη και μέσα στον υπολογισμό για την επόμενη επταετία στο πολιτισμικό οικονομικό πλαίσιο που η Επιτροπή υποστηρίζει πω 25% του προπολογισμού ε, να πρέπει να πάει σε περιβαλλοντικές ε, δράσεις, δηλαδή 323 εκατομμύρια ευρώ ε, σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα για τις υποδομές, ε, για την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία, την γεωργία. 25% επίσης από το ορίζον θα πρέπει να στοχεύουν σε στόχους περιβαλλοντικούς, 50 δισεκατομμύρια για το κλίμα, την ε, κινητικότητα, τεχνολογία, ορίζων Ευρώπη θα ε, πρέπει να στοχεύει σε φύσεις πόλεις, ουδέτερες ε, κλιματικά και να εξασφαλίσει 5 με 10 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση. Επιπλέον προτείνουμε ένα 30% των επενδύσεων στο InvestEU που δια, ε, που ακολουθεί το σχέδιο Juncker να ε, πάνε αντίστοιχα σε περιβαλλοντικές δράσεις. Με 5 δισεκατομμύρια ευρώ μπορούμε να έχουμε δράσεις ανάπτυξη ικανοτήτων για συνεργασίες ΣΔΙΤ και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας. Οι προτάσεις μας είναι φιλόδοξες, είναι προτάσεις όμως που μπορούν να επιτευχθούν και μπορούν να δημιουργήσουν το πιο σημαντικό επιπλέον χρηματοδοτικές δυνατότητες για τις πόλεις, για τους πολίτες, για την προσαρμογή αλλά και τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών. Και θα ήθελα ολοκληρώνοντα να σας ε, συγχαρώ για τη δουλειά που κάνετε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά, η σημερινή σας συζήτηση και ο αναλογισμός μας επιτρέπεται με τις προσπάθειές σας να εντοπίσουμε τις καταλληλότερες δράσεις και τη δουλειά που χρειάζεται να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υποστηρίξουμε τις δικές σας δράσεις. Ταυτόχρονα βέβαια αναγνωρίζοντας και τις ε, διαφορές και τους παράγοντες τους καθοριστικούς στις περιοχές χωριστά την κάθε της καθεμίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημαντική σας συμβολή μέχρι τώρα και στο μέλλον σε αυτή τη σημαντική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire, pour ce tour d'horizon euh, très concret et très complet. Et nous allons maintenant Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ακούσουμε τους ε, συναδέλφους της Επιτροπής των Περιφερειών. Πολλοί έχουν στήσει το λόγο. Κλείνω προσωρινά τον κατάλογο για τις παρεμβάσεις σας, ε, παρακαλώντας σας να τηρήσετε αυστηρά το χρόνο, ιδάλλως κινδυνεύουμε να βγούμε εκτός προγράμματος. Γι' αυτό και ζητώ την ε, κατανόησή σας. Αν τυχόν χρειάζεται να σας περιορίσω. Πολιτικές ομάδες πρώτα. Πρώτος αντιπρόεδρος. Κύριος Ρίμπανη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κανιέτε, Σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας δείτε για να μας μιλήσετε για αυτά τα σημαντικά θέματα. Η έκθεση πρωτοβουλίας που, η πρωτοβουλίας που κατάρτισα εκ μέρους ομάδας μου με ενδιαφέρει, θα ήθελα να σας την αναφέρω, καθώς προέρχομαι από μια περιοχή που έχει ορίσει δικούς της κλιματικούς ε, στόχους και θα ήθελα να συγχαρώ εσάς αλλά και το προσωπικό σας η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ρόλο ηγετικό στην προάσπιση του κλίματος και την αντιμετώπιση της ενεργειακής μετάβασης. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή συζήτηση. Χρόνια τώρα αντιμετωπίζουμε ε, έκτακτα και ακραία καιρικά φαινόμενα με κυκλώνες ακόμα που εκδηλώνονται στην κεντρική Ευρώπη και είναι σαφές το αναγνωρίζει και ο πολίτης ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως ε, μέχρι τώρα. Ε, άρα λοιπόν πρέπει να περάσουμε σε μια παραγωγή βιώσιμη και ένα σύστημα βιώσιμης κατανάλωσης. Χρόνια τώρα κάνω αυτή τη δουλειά ε, και ασχολούμαι με τα θέματα αυτά εκ μέρους της ε, πόλης που εκπροσωπώ και θέλω να ρωτήσω το εξή. Στόχοι 2030. Αυτοί πρέπει σε εθνικό επίπεδο να μεταφράζονται σε συγκεκριμένες δράσεις. Άρα πρέπει να υπάρχουν συστήματα προσαρμογής στις ενεργειακές πηγές που να υπηρετούν το στόχο του ορίζοντα 2030, λαμβάνοντας υπόψη του στόχους και του 2050. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να πείσουμε πολίτη και επιχείρηση ιδιωτική για το μοντέλο αυτό ανάπτυξης. Πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα αγοράς ώστε να προσαρμοστούμε πιο γρήγορα στις ε, ανάγκες, στις επιταγές της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, Χρειάζεται παρέμβαση για να τηρηθούν αυτοί οι στόχοι, να υπάρχουν εγγύησεις δηλαδή, να υπάρχει ο σχεδιασμός οριμοτομικός, η ενεργειακή παραγωγή, οι διαγωνισμοί για τις προμήθειες, για τις μεταφορές, όλα αυτά πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις επιταγές της κλιματικής αλλαγής. Έτσι λοιπόν, από μας ε, πρέπει νομίζω να έρθει ένα μήνυμα γιατί μπορούμε με την εμπειρία που έχουμε να δώσουμε και ένα παράδειγμα για μετα, ε, μετάβαση και προσαρμογή. Πρέπει τα κράτη-μέλη να ακούσουν προσεκτικά αυτά που έχουμε να πούμε εμείς για αυτά τα ολοκληρωμένα ενεργειακά σχέδια τα οποία έχουν κέρια σημασία για μια ανανέωση στον τομέα της, ε, του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής. Πρόκειται για μια πρόκληση μεγάλη παγκόσμια. Στηριζόμαστε βέβαια. Παρακαλώ, λέει ο πρόεδρο, να τελειώσετε. Δεν έχω άλλο περιθώριο να σα αφήσω το χρόνο. Το έχετε εξαντλήσει. Και τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Εμιλιάνο. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο για την παρουσία του εδώ σε αυτό το κρίσιμο σημείο χρονικά, όχι μόνο για τον πολίτη μας, αλλά και, γενικότερα, και ειδικότερα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωση, η κλιματική αλλαγή καθημερινά μας ε, επιδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σε κάθε περιφέρεια της Ευρώπης και πόσο απαραίτητο είναι να εισαχθούν κατεπηγόντα μέτρα. Είναι τεράστια η πρόκληση, πρέπει να εντοπίσουμε νέα παραγωγικά συστήματα, νέα συστήματα κατανάλωσης και να ζήσουμε πράγματι μέσα στα όρια των πόρων που διαθέτει ο, ο πλανήτης μας έτσι ώστε να αφήσουμε ε, ένα υγιή πλανήτη στο, στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ήταν πολύ σημαντικές ε, οι πρωτοβουλίες και τα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις συμφωνίες των Παρισίων με την υιοθε... και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα με την υιοθέτηση των στόχων ε, της βιώσιμης ανάπτυξης και η αντίληψη ότι εμείς στην Ευρώπη πρέπει να, να βγούμε στην πρωτοκαθεδρία, στην πρωτοπορία της αλλαγής ε, γιατί έχουμε και την ιστορική ευθύνη που μας υποχρεώνει σε αυτό. Κύριε Επίτροπε θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δουλειά σας, για την ε, διάβγεια της ε, δράσης σας που μας οδήγησε στον δρόμο αυτό. Βέβαια είναι μεγάλη η πρόκληση και ε, στο μέλλον πρέπει να παραμείνουμε ε, αποτελεσματικοί αλλά και να συνεχίσουμε με μέτρα τα οποία θα είναι περιεκτικά, δεν θα αποκλείουν κανέναν αλλά δεν είναι και ισότιμα εν ώψη των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Εμείς σοσιαλιστές και προοδευτικοί δεν λησμονούμε μια σημαντική διάσταση αυτού του αγώνα. Πρέπει ο αγώνας λοιπόν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του περιορισμού των συνεπειών της να συνοδεύεται και από μια, ένα αγώνα για κοινωνική ε, ισότητα και δικαιοσύνη που δεν θα επιτρέψει να αποκλειστεί κανείς ε, από την πρόοδο στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορέσει να καταλήξει μια ε, ομόφωνη απόφαση για τα ζητήματα αυτά και ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει τις ε, διαφωνίες, τις διαφορές επόψεων και ελπίζω επίσης ότι οι γείτονες και οι σύμμαχοι με τις ΗΠΑ Αμερικής σε θα μπορέσουν να βρουν μια απάντηση σε ε, προβλήματα ήδη Υπάρχει ένα Climate Action Now Act, ένας νόμος δηλαδή δράση ε, τώρα για το κλίμα που υιοθέτησε η Βουλή των Αντιπροσώπων πρόσφατα, και με την οποία καλείται ο πρόεδρος ε, Τραμπ να ε, προσχωρήσει και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις των Παρισίων. Ε, είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την, την Επιτροπή των Περιφερειών και καλούμαστε να δώσουμε σημαντική συμβολή με την, διάδοση, με την διάχυση μιας συνειδητοποίησης, μιας κοινή συνειδητοποίησης της σημασίας αυτών των πολιτικών. Ο, ε, η γνωμοδότηση που θα συστήσουμε και που έχω εγώ συντάξει με την κυρία Κατατιούτο ε, έχει θεμελιώδη ε, σημασία. Πιστεύω ιδιαίτερα για τις χώρες που ε, βλέπουν πως χρειάζεται ενεργειακή ισότητα που θα λαμβάνει υπόψη και την πολιτική προστασία του περιβάλλοντος χωρίς όμως να την μετατρέπει σε ένα ε, στοιχείο επιπλέον ανταγωνιστικότητας και ανταγωνισμού. Και θα ήθελα σε θεσμικό επίπεδο τώρα να εκφράσω την ελπίδα πως η Επιτροπή και ολοκληρώνοντας την παρούσα θητεία αλλά και η προσεχής που θα αναλάβει να μπορέσει να, δώσει την ίδια, να προσδώσει την ίδια προσοχή ουσιώδη και γνήσια που εσείς επιδείξατε στα θέματα αυτά της ενέργειας. ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Τι ετάρι, παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ευρωεκλογέ κατέδειξαν ότι υπάρχει ευρεία στήριξη από τον πληθυσμό για την ενεργειακή μετάβαση. Αλλά δεν φαίνεται ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν κατανοήσει αυτή την επιθυμία. Τέσσερα κράτη-μέλη, όπως ακούσαμε, παρεμπόδισαν τη λήψη αποφάσεων για μια στρατηγική για το κλίμα μέχρι το 2050. Εμείς οι τοπικοί και περιφερειακοί εκλεγμένοι πρέπει να εργαστούμε περισσότερο γιατί είναι μια καθημερινή πρόκληση η κλιματική αλλαγή και πρέπει ήδη να επενδύσουμε στις αναγκαίες υποδομές. Γι' αυτό το ερώτημα τι θέλουμε όντως να γίνει κάτι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να περιμένουμε. Πρέπει να βγούμε από μια κατάσταση αδράνειας λόγω της τάσης κάποιων κρατών μελών. Γιατί δεν μας δίδεται ήδη σε εμά ε, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές το ρόλο που θα μπορούσαμε να παίξουμε. Αυτό το ερώτημα θέλω να απευθύνω και σε εσά αγαπητέ κύριε Επιτροπέ. Η συνάντηση κορυφής στο Νέα Υόρκη και η COP25 στην Χιλή επίκενται. αλλά δεν έχουμε ακόμη δεσμεύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση Άρα δεν θα έχουμε και μια σωστή διαπραγματευτική θέση. Δεν θα έχουμε διαπραγματευτική εντολή επιπλέον. Περιορίστηκε και η εντολή που θα δώσουμε στην αντιπροσωπεία μας. Πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσεις μας να δράσουν και η αντιπροσωπεία μας να λάβει την αναγκαία εντολή και να ε, συμπεριλαμβάνει και εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Είναι αναγκαία όλα αυτά για να μπορέσουμε πραγματικά να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κούπο. Πού πάμε λοιπόν. Με τις οικονομήσεις άνθρακα παντού στον κόσμο και με τις εθνικές συμβολές θα έχουμε μια αύξηση 3,5 βαθμών στην παγκόσμια θερμοκρασία. Σημαίνει αυτό πλημμύρε στις πόλεις μας. Ένα μεγάλο τμήμα των εδαφών μας ε, θα γίνει έρημο. Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε σοδιές και θα υπάρξει μαζική μετανάστευση. Θα αποτύχουμε. Δεν είμαστε επαρκώς φιλόδοξοι για να κάνουμε αυτό που είναι απόλυτα αναγκαίο. Δεν είμαστε επαρκώς φιλόδοξοι ούτω ώστε αυτά που ζητούν τα εκατομμύρια ατόμων που απαιτούν περισσότερα. Η διαδικασία COP προβλέπει όλο και αυξανόμενο ρόλο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Εμείς ως Επιτροπή Περιφερειών θέλουμε οι συμβολές να καθορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Αυτό το στηρίζει και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οργανισμοί παντού στον κόσμο. Και υπεντεύχθη κάποια πρόοδος. Τώρα έχουμε έχουμε την λήψη υπόψη των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών. Αλλά η δική μου τοπική αρχή δεν έχει έρθει κανεί σε επαφή μαζί μα από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Φαίνεται έχουν άλλα πράγματα να κάνουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πολλά γίνονται από τις τοπικές αρχές που κηρύσουν ότι υπάρχει κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που λένε ότι οι στόχοι του παγκοσμίου, του διεθνούς ε, πάνελ για την κλιματική αλλαγή πρέπει να υλοποιηθούν. Δεν έχουμε όμως γίνει εκεί στη, στον Ρωμανό Βασίλειο αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ε, δεινόσαυρους ως ηγέτες γιατί θα εξαφανιστούμε όπως οι δεινόσαυροι τελικά. Ευχαριστώ. Βλάζακ. Ευχαριστώ πολύ να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να ασχοληθώ με την ενεργειακή μετάβαση σε περιφέρειες που ε, εξαρτώνται από ρητά καύσιμα. Χαίρομαι που λαμβάνουμε χρηματοδοτική βοήθεια από την Ένωση για τη μετάβαση αυτή. Για παράδειγμα, έχουμε τις ε, περιφερειακές πλατφόρμες για τον άνθρακα, γιατί μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε για να ξεκινήσουν πολύ σημαντικά πιλωτικά προγράμματα σε διάφορα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Τσεχική Δημοκρατία, αλλά και η Πολωνία και η Σλοβακία. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί και ότι θα στηριχθεί με την επαρκή χρηματοδότηση. Λόγω του τρόπου με τον οποίο ε, παράγουμε ενέργεια, χρειαζόμαστε βοήθεια, ιδιαίτερα στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξετάζοντα τι προοπτικέ αυτέ τι περιοχέ οικονομική ανάπτυξη, διαπιστώνουμε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο ο άνθρακα. Ήταν όντω ο κινητήρα των οικονομιών μα. Όπω έγινε και στη Δυτική Ευρώπη κατά τη βιομηχανική επανάσταση για διάφορους αιώνες στην Όστραβα στην ε, βορειοανατολική Τσεχική Δημοκρατία, στη Βαλονία, στην Βόρεια Αγγλία. Ο άνθρακας ήταν ε, το πρώτο αγαθό και ο λιθάνθρακας υψηλή ποιότητας ήταν ε, ακόμη καλύτερος. Στον 20ο όμως αιώνα μειώθηκε η κατανάλωση άνθρακα και αυτό δημιούργησε υψηλή ανεργία και κοινωνικά προβλήματα. Ο άνθρακας είχε βοηθήσει τις περιοχές αυτές να γίνουν η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά όταν καταργήθηκε η εξόριξή του, οι περιοχές αυτές καθυστέρησαν πολύ και υπέστησαν τις συνέπειες. Βεβαίως βελτιώθηκε στην Όστραβα το Σαλεγουά και το Μάντσεστερ, βελτιώθηκε η ποιότητα του αέρα, αλλά καταστράφηκε η απασχόληση. Ο Winston Churchill είπε ότι όσοι δεν ε, μαθαίνουν από την ιστορία είναι καταδικασμένοι να την παραλαμβάνουν. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε, γιατί στην Ένωση ακόμη έχουμε 240.000 θέσει εργασία, απευθεία, σχετιζόμενε με την εξόριξη άνθρακα. Αν δεν μάθουμε από την ιστορία, αυτέ τι θέσει εργασία που οι περισσότερε από αυτέ είναι σε περιφέρειες χαμηλού ΑΕΠ θα χαθούν. Αν κλείσουμε πριν το 2030 τα ανθρακοριχεία θα χάσουμε βάση εκτιμήσεων 160.000 θέσει Χάριστε χάρη στην αναδιάρθρωση της οικονομίας και την ε, οικονομική βοήθεια για τις βασικές ε, επιχειρήσεις σε αυτή την περιοχή τα καταφέραμε μέχρι τώρα ελπίζω να κάνουμε περισσότερο ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μάρκου Μάρκουλα τώρα ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι καταρχάς ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε με το περιφερειακό επίπεδο και το τονίζετε. Και εμείς ακούσαμε και από τον κύριο Κατάινεν κάτι ε, παρόμοιο όταν αναφέρθηκε στην βιώσιμη ανάπτυξη ότι συμμετέχουμε και εμείς εκεί. Ένα στοιχείο που τονίσατε είναι ότι δεν υπήρχε αυτή η τοπική και η περιφερειακή διάσταση μέχρι τώρα. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να είναι παρόντε κατά τι διαπραγματεύσει και κατά τη λήψη αποφάσεων. Όταν θα αποφασιστεί ακριβώ τι θα γίνει για το κλιματικό θέμα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σα. Είμαστε 350 τοπικά εκλεγμένοι και θα είχαμε όλη τη δυνατότητα να δώσουμε ευρύτερη στήριξη και να βελτιώσουμε την εφαρμογή των μέτρων και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Να είμαστε ένα πρότυπο για ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτω ώστε να δώσουμε σε όλου μα συμπολίτε τη βεβαιότητα ότι συμμετέχουν. Έτσι θα είμαστε υπόδειγμα και παγκόσμια. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε όντω να προωθήσουμε του στόχου μα. Σήμερα το πρωί, εδώ εμείς στην Επιτροπή μας ακούσαμε διάφορους ε, συναδέλφους, κάναμε ανταλλαγή απόψεων, συζητήσαμε τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε και περισσότερα, ούτω ώστε να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι όλα τα κράτη-μέλη θα εκπονήσουν εθνικά προγράμματα ε, ενεργειακής μετάβασης και αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Αλλά αν δεν προβλέπονται κυρώσεις συγκεκριμένα μέτρα και εφαρμογή με αποφάσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν ο καθένας μας, στην πόλη μας, στην περιφερειά μας, να προσαρμόσουμε τα προγράμματα αυτά και μετά να τα ε, αποστείλουμε τις αποφάσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις ε, κυβερνήσεις, ούτως ώστε να ασκηθεί πίεση και κάποια άλλα ζητήματα. Σήμερα δημοσιεύεται ένα άρθρο μου σε μια μεγάλη φινλανδική εφημερίδα μαζί με τον ε, κύριο Λάπαλάινεν είπαμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε καλές εταιρικές σχέσεις και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Χρειαζόμαστε να ξεκινάει από τις κοινότητες η καινοτομία αλλά και η κυβέρνησή μας πρέπει να καταλάβει τι σημαίνουν όλα αυτά. Στόχος μας πρέπει να είναι ότι το 2035 η Φιλανδία πρέπει να είναι ε, ουδέτερη από πλευράς ε, εκπομπών άνθρακα. Αλλά θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο αυστηροί. Γιατί πολλά ακόμη πρέπει να επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμη 16 ομιλητές λέει ο πρόεδρο. Ένα λεπτό καθένα και θα είμαι αυστηρό. γιατί αλλιώ ε, θα καθυστερήσουμε τις περαιτέρω εργασίες μας. Λοιπόν, η κυρία Τούτε είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ που δείτε το λόγο. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ τον ε, χρόνο αγόρευση. Συζητούμε εδώ την ενεργειακή μετάβαση, τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει και αυτό μου υπενθυμίζει μάλλον μου θυμίζει ένα ε, τρένο που μπροστά έχει την ε, μηχανή και πίσω έχει ε, τους, τα βαγόνια που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον, την ταχύτητα της μηχανής και έτσι κάποια μένουν πίσω. Αυτό μπορεί να ισχύει και για 50 εκατομμύρια Ευρωπαίους για τους οποίους ενεργειακή φτώχεια σημαίνει ότι δυσκολεύονται να πληρώσουν τη θέρμανση το χειμώνα. Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι φιλόδοξα, να έχουν όνειρα, Η εσύ είναι κάτι σημαντικό, η εξέβρεση μιας πολύ καλής δουλειάς. Θέλουμε να τα δούμε αστροφυσικούς ε, μια μέρα, αλλά αν δεν μπορούν να διαβάσουν σε ένα δωμάτιο ζεστό και να φάνε ένα πιάτο φαγητό το βράδυ, πώς θα τα πετύχουν όλα αυτά τα παιδιά μας. Και αυτό είναι πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και παντού. Διακόπτεται η ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ήταν εμπνευσμένο ο λόγος σα. Εγώ θα εστιάσω στα δύο σημαντικότερα για μένα ε, σημεία σε αυτό το μοναδικό λεπτό που έχω στη διάθεσή Το ρόλο της τοπικής ε, ε, και περιφερειακής αρχής που είναι κοντά στους πολίτες πρέπει να έχουν ε, ε, να οικειοποιηθούν ε, την προστασία του κλίματος. Έχουμε από το ΛΟΤΣ μια από τις 41 περιφέρειες που εξαρτάται από τον άνθρακα, από τα, τα κάψιμα και πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Πρέπει να μειωθούν εκπομπές, ιδίως ε, το 2050. Παραγωγή λιγνίτη επίσης πρέπει να μειωθεί στο Μπουρχάτοφ μια άλλη περιοχή. Τεράστια πρόκληση, διότι το μέρος αυτό της Πολωνίας βασίζεται στη βιομηχανία αυτή. Μιλάμε για πάνω από 4 δις ευρώ ε, για ενίσχυση αυτής της περιφέρειας και αυτά τα χρήματα πρέπει να τα βρούμε. Διακόπτεται και αυτός ο Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Είμαι από την Κρόσνα Μπόκα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη Ρουμανία στην Τρανσιλβανία, στο κέντρο τη Τρανσιλβανία. Είμαι δήμαρχο εκεί. Εμεί προσπαθούμε να πετύχουμε την πράσινη κινητικότητα μέχρι το 2025. Για παράδειγμα, θα έχουμε ηλεκτρικές δημόσιες συγκοινωνίες Θέλουμε κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2051, ένα όραμα στο οποίο συμμερίζομαι. Το θέμα δεν είναι μόνο πώ θα πετύχουμε όμω αυτό το στόχο. Έχω δύο σχόλια επ' αυτού. Πρώτον, νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσουμε την επικοινωνία μα με του πολίτε. Διότι πρέπει να είναι και οι πολίτε μαζί ε, σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητούν οι ελίτ μόνο. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση άλλο να ε, επικοινωνούμε προς τους πολίτες ε, και άλλο μαζί με τους πολίτες ε, γιατί παραδείγματο χάρη μπορούμε το κάψιμο να το δεχθούμε όχι όμως να τους φέρει ρήπανση οι συμπράξεις δημόσια τομέα είναι κάτι σημαντικό και από όλα άλλα μέτρα το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε La parole maintenant notre Τώρα, κύριε Χωνή. Πρόεδρε, Επίτροπε Καρνιέτε. Καλωσορίζω την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα καθαρό πλανήτη για όλους. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2050 με την καταπολέμηση της κλιματικής αναγής, ε, αλλαγής ακόμη πιο εντατική. Είμαι πεπισμένη πως οι πόλεις μας ε, και οι περιφέρειές μας χρειάζονται μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα μας προσφέρει ένα φιλόδοξο πλαίσιο και θα δίνει ε, κατευθύνσεις και μέσα όμως για την μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει τον στόχο, να επιτύχει τον στόχο της ε, ουδετερότητας ως προς τα αέρια θερμοκηπίου να τον ε, επιδιώξει πολύ πιο εντατικά στο 2050. Δυστυχώς δεν συμφώνησαν οι Υπουργοί. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει για την εκμυδένιση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό πρέπει να γίνει κατά τρόπο κοινωνικός ε, αποδεκτό. Άλμιγκερ Μίλγκερ παρακαλώ. Κύριε Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που είχαμε την, έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητούμε το θέμα αυτό, που είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ, ιδιαίτερα τους νέους στην ε, δική μου την ιδιαίτερη πατρίδα, μια περιφέρεια της Αυστρίας με 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, με πολύ έντονη παρουσία και της ερευνητικής δραστηριότητας ε, και ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες τεχνολογίες στην ερευνητική μας δραστηριότητα. Ε, έχουμε λοιπόν μια μικρή δυνατότητα με 2,5 εκατομμύρια ε, πολίτες, ε, μικρή δυνατότητα να συγκρατήσουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά έχουμε πολλά να προσφέρουμε ως μέσα χάρη στην έρευνά μας. 550 εκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα, ε, δηλαδή 40% περισσότερο από όσο θα μπορούσε η δική μου η περιφέρεια να ε, εκπέμψη μπορούμε να εξοικονομούμε χάρη στις μεθόδους που εφευρίσκονται στην ε, περιοχή μου. Και επίσης, ε, και άρα μπορεί μια μικρή περιοχή να κάνει πάρα πολλά για τον πλανήτη επίσης. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη και η κλιματική, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής μπορούν να πηγαίνουν χέρι-χέρι και να μην είναι ε, στους αντίποδες. Μπορούν να συνδυαστούν. Ευχαριστώ πολύ. Έχει περάσει ο χρόνος σας λέει ο Πρόεδρος και τώρα ακούμε τον κύριο Ρώση. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκφράζω και εγώ την ικανοποίησή μου για τις ε, πρόοδους ε, στην κυκλική οικονομία. Πολλές ε, περιφέρειες ε, εμπνεύστηκαν ε, από τους κανονισμούς και τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλές φορές προλαμβάνοντας τις επιταγές τους. Παραδείγματι το Σκάνι ως περιφέρεια έχει μέχρι το 2030 το στόχο της αγωγής της πλήρους ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων αλλά και την τον απόλυτο διαχωρισμό αποβλήτων για την ανακύκλωση. Μέχρι το 2050 μπορούμε να έχουμε ε, υλοποιήσει το στόχο της ουδετερότητας ως προς το διοξίδιο, την ε, κατάργηση του πλαστικού μίας χρήσεως, όλα αυτά τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε μόνο εφόσον συνεργαστούν και οι πολίτες με μια μεγάλη όθηση και ιδιαίτερη πίεση από τις τοπικές αρχές, από τους, τα κοινωνικά κινήματα και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις μας έχουν βοηθήσει στους στόχους αυτούς και θέλουμε η φωνή μας να ακουστεί πιο δυνατά ακόμη διότι πιστεύω ότι ο πολίτης πάνω απ' όλα ο νέος ε, τα θέματα του περιβάλλοντος είναι πολύ πιο μπροστά και από την πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Ε, πέρασε και ο χρόνος σα. Μάρκης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω πως οι πιο ευάλωτες περιοχές ε, και από τις αστικές, τις απομακρυσμένες ή τις νησιωτικές εκείνες είναι οι ορεινές περιοχές, οι οποίες μάλιστα προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες στις παιδιάδες και στα αστικά κέντρα. Είναι από θέματα υδάτων, είναι θεματοφύλακες των, ε, της χλωρίδας και της πανίδας, καθαρίζουν το περιβάλλον και η δική μας η μικρή μικρή περιοχή της Βάλεντα λαός έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για τις μερικές εκατοντάδες χιλιάδων των κατοίκων της αλλά για όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης 500 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν μια περιοχή η οποία πρέπει να προστατευθεί και ως προς το λιώσιμο των πάγων και ως προς τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ε, εμεί ω ομάδα λέμε πως δεν είναι δυνατόν μόνη της να επιβαρύνεται με το κόστος περιορισμού των ε, κινδύνων ή μεγιστοποίησης των ωφελών η ε, περιοχή μας πιστεύω ότι ότι ακόμα και με τα κονδύλια που μπορεί να προβλέπονται δεν αρκούν αυτά για να υλοποιηθούν σε ολοκληρωμένο τρόπο οι στρατηγικές μας και τα σχέδιά μας και πιστεύω ότι θα πρέπει τα υψίπεδα εκείνα και οι ορεινές περιοχές να έχουν στο δυνατόν καλύτερη διακήρυξη. Ο πρόεδρος διακόπτει και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λίμαν. Αγαπητοί συνάδελφοι. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Έχουμε να κάνουμε με τις ε, εξελίξεις στην τεχνολογία, με τα πιο ε, εξελιγμένα, προηγμένα, μοντέρνα συστήματα εκμετάλλευσης του λιγνίτη. Παρόλα αυτά όμως δεν θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε μετά το 2050 και θα χάσουμε 350.000 θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες θέσεις βιομηχανικής παραγωγής που θα οδηγήσουν και σε μια διαρθρωτική ε, αλλαγή, σε ένα ρήγμα στρατιωτικό. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει να υπάρξει μια αντίστοιχη ε, επιτροπή με εκπροσώπους των κοινοτήτων, των περιφερειών της Ομοσπονδιακής ε, Κυβέρνησης για να βοηθήσουν στην ε, αντιμετώπιση των διεθνωτικών αυτών μεταλλάξεων. Μέσα από στοχευμένες λοιπόν επενδύσεις υποδομές, σε υποδομές, εκπαίδευση και νοτομία μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερες νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας για τη βιομηχανική παραγωγή που θα συγκρατήσουν και τους πολίτες μας στις περιοχές μας. Ελπίζω πράγματι να έχουμε και ένα πλαίσιο υποστήριξη ευρωπαϊκό επίπεδο με, την ενίσ, με τις ενισχύσεις και τα κονδύλια που χρειάζονται για τις 51 περιοχές ε, ε, παραγωγής λιγνίτη που δεν πρέπει να εγκαταλευτούν στη μία. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Έχει λήξει ο χρόνος σας, ο κύριος Ζήγελ. η κλιματική αλλαγή δεν, δεν μεγάλη σημασία μόνο και μόνο επειδή κατεβαίνουν τα παιδιά στους δρόμους κάθε Παρασκευή με το Fridays for Future. Όχι, πρέπει να χαιρετήσουμε εδώ τις μεγάλες αλλαγές και τις προτάσεις, τη δυνατότητα για εξασφάλιση στόχων που πολλές φορές καλούνται να ε, αντιμετωπίσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις τους. Λυσμονούνται πολλές φορές και σε αυτό θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να προσφέρουμε με βάση την επικουρικότητα και αυτό θα πρέπει να γίνει ζώσα πραγματικότητα. Η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί με τα hubs για την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού δικαίου στις διάφορες περιφέρειες να συμβάλλει με την επαλήθευση της επικουρικότητας και τα περιφερειακά hubs μπορεί να αξιοποιηθεί και η δουλειά της Επιτροπής των Περιφερειών στο κλίμα και την ενέργεια, στις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια μπορούμε πολλά να ε, προσφέρουμε μέσα από τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές και βέβαια απαιτούμε και εμείς να λαμβανόμαστε με σοβαρότητα υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Κάλα Μπουίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να συγχαρώ την Επιτροπή για τις προσπάθειες που κάνει για να γίνουν πραγματικότητα οι δεσμεύσεις, ε, οι τόσο ουσιώδεις που έχουν να κάνουν την κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα με τους στόχους για το 2050 αλλά είναι επίσης προφανές ότι οι περιφέρειες έχουν ουσιώδη ρόλο να παίξουν και ιδιαίτερα σε χώρες που είναι τόσο σημαντικές όπως η Ισπανία και χρειαζόμαστε την επαρκή χρηματοδότηση γι' αυτό για να μετοπίσουμε τεράστιες προκλήσεις και για να προλάβουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις να μην ε, ξεχάσουμε κανένα δηλαδή Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή μέσω τη ενεργειακή μετάβαση. Και δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνη ή προστασία του περιβάλλοντο. Είναι θέμα επιβίωση, ασφάλεια για του συμπολίτε μα. Υπάρχουν ε, περιφέρειες που είναι πολύ ευάλωτε, όπω είναι συνολικά η Μεσόγειο. Εκεί έχουμε πολύ ακραία φαινόμενα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Ταραγώνα υπάρχει μια τρομερή πυρκαγιά και θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τους πολίτες που έχουν θυγεί και με τις δυνάμεις που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά. Και επίσης πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη διαδικασία μετάβαση να δημιουργήσει περισσότερη φτώχεια. Ευχαριστώ πολύ. Σύρπα Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι από το ΕΛΚ κύριε Κανιέτε και είμαι εισηγήτρια για τα ενεργειακά και κλιματικά θέματα και είμαι δημοτική σύμβουλος από το ΕΣΠΟ. Ο κύριος Μάρκουλα αναφέρθηκε ήδη στο Δήμο μου του ΕΣΠΟ. Λοιπόν, να τονίσω τα εξή. Πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση για την κλιματική αλλαγή να προσαρμοστούν οι στόχοι της Ένωσης στους στόχους 2030 και στη Συμφωνία των Παρισιών, οι περιφέρειες και οι πόλεις. Είναι αρμόδιες για 90% των μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ένωση λοιπόν σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές θα επιτύχει του στόχου. Χρειαζόμαστε πράσινε και γαλάζιε επενδύσει και καινοτομία. Θέλουμε το 30% να ληφθεί υπόψη για τις ε, καινοτόμες ε, επενδύσεις. Ο συνάδελφος Μπράτισλαβ Κλίνκα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ την Επιτροπή Περιφερειών και όλους τους συζητητές και συναδέλφους που συνέβαλαν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσω των γνωμονωτήσεών μας. Τονίζω τη σημασία του θέματος αυτού για τις περιφέρειες. Στην ε, Τσεχία οι διαδικασίες είναι συγκεντρωτικές. Η κυβέρνηση αποφασίζει για το μέλλον των μεμονωμένων περιφερειών ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους. Και αυτό δεν μας επιτρέπει να επιτύχουμε τους στόχου της Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την κυκλική οικονομία, την εισαγωγή ανανεωσίμων και άλλα θέματα. Και έτσι δεν αντιμετωπίζεται το θέμα. Δεν προωθούμε τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Εάν δεν υπάρξει λογική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Και ελπίζω ότι αν συνεργαστούμε σωστά θα αλλάξουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Καραγιάννης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρκετοί ομιλητέ και αρμόδιοι επίτροποι έρχονται στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και μα συμβουλεύουν πώ να σεβόμαστε το περιβάλλον, η αποφυγή τη περιβαλλοντική καταστροφή, τη κλιματική αλλαγή και την ανακύκλωση και για να σεβόμαστε την εφαρμογή της συμφωνίας του παρισιού για την κλιματική αλλαγή την οποία παρεμπιπτόντως κάποιες χώρες δεν σέβονται ούτε εφαρμόζουν. όμως κύριε πρόεδρε δεν είμαστε εμείς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που μολύνουν τους ωκεανούς άλλων χωρών ιδιαίτερα στην νοτιοανατολική ασία με τα απόβλητα που εξάγουμε δηλαδή τα πλαστικά δεν είμαστε εμεί οι τοπικέ αρχέ που εξάγουμε τα ρηπογόνα παλιά πετρελοκίνητα αυτοκίνητα και τα στέλνουμε στα βαλκάνια και στη μέση ανατολή. είναι οι χώρε μα, είναι οι χώρε μέλη. άρα κύριε επίτροπε θέλουμε καθαρό περιβάλλον στην ευρώπη στην ευρωπαϊκή ένωση αλλά μολυσμένο περιβάλλον σε άλλου ωκεανού και σε άλλε υπήρους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κοιτάξτε, να αναφέρω κάτι που δεν αναφέρθηκε. Αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές, τι θα γίνει με τα πυρηνικά εργοστάσια. Επισήμως θεωρείται ότι είναι μηδενικών εκπομπών. Όμως είναι τμήμα μιας αλυσίδας εφοδιασμού που, που ξεκινάει από τα ορυχεία ουρανίου. Και στην άλλη άκρη φυσικά είναι ε, η, η αντιμετώπιση των πυρηνικών αποβλήτων. Εδώ παίζουν ρόλο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Γιατί τα θέματα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο στην κοινωνικονομική ανάπτυξη. Πολλοί από εμά έχουμε στις περιφέρειές μας ε, τέτοια πυρηνικά εργοστάσια. Άρα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πώ θα διαχειριστούμε τα απόβλητα, πώ θα διαχειριστούμε μακροχρόνια την ε, ε, αποσυναρμολόγηση αυτών των ίδιων των εργοστασίων. Υπάρχει μια ομάδα εργασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων που προσπαθεί να προβλέψει τι ε, επιπτώσει θα ε, προκύψουν. Είμαι από μια μικρή πόλη όπου θέλουν να ξεκινήσουν ένα νέο μεταλλείο ουρανίου και ένα χώρο για εναπόθεση των αποβλήτων. Τι θα γίνει. Πρόεδρο, όπως συζητάμε την ενεργειακή μετάβαση, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ε, πρέπει να έχουμε τοπική προσέγγιση. Εγώ είμαι μέλος ε, της συνέλευσης του Λονδίνου. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ε, στην πολιτική μας για τις συγκοινωνίες. Έτσι θα βελτιώσουμε την κατάσταση παντού στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσει πρέπει να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία δίνει νομική βεβαιότητα χωρί να δημιουργεί περισσότερη γραφειοκρατία που πνίγει την καινοτομία. Οι κυβερνήσει πρέπει να δημιουργήσουν ένα γενικό πλαίσιο και να επιτρέψουν στι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ να υιοθετούν ταχύτερα μέτρα για να προσαρμόζονται στην ε, τεχνολογική εξέλιξη. Έτσι οι επιχειρήσει θα καινοτομούν μέσω ενό ελαφρού ρυθμιστικού πλαισίου. Η ενεργειακή μετάβαση και η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής είναι ένα τομέα όπου το Ηνωμένο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσουν να συνεργαστούν ακόμη και όταν τον Οκτώβριο θα αποχωρήσουμε. Και προσβλέπω στη συνέχιση του διαλόγου για αυτό και άλλα σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταίο ομιλητή, ο, ο συνάδελφο Ραφαέλε Κατανέο. Κύριε Επίτροπε, ω υπεύθυνο για, για το περιβάλλον και το κλίμα στην Λομβαρδία, στην περιφερειά μου. Μπορώ να πω ότι γνωρίζω καλά τα ζητήματα. Έχουμε τριπλάσιο αντίκτυπο στις δράσεις μας εμείς οι περιφέρειες από ότι οι κεντρικές κυβερνήσεις και γι' αυτό ζητώ την ενίσχυση και της υποστήριξη που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα, η ενεργειακή των κτηρίων που ήδη υπάρχουν, η ενέργεια που θα κοστίζει λιγότερο, που θα έχει μηδενικές εκπομπές, μπορεί να είναι μόνο η ενέργεια που δεν καταναλώνεται και έτσι χρειάζεται μια υποστήριξη πολιτικών που θα οδηγήσουν όχι σε εκμηδενισμό αλλά σε ε, μείωση στο δυνατόν ή στη βελτίωση στο έπακρο τη ενεργειακή αποδοτικότητα για να γνωρίζει και η κάθε οικογένεια τι προσφέρεται και για να ενισχυθούν οι τοπικέ και περιφερειακέ πολιτικέ ε, προ το στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση ενέργεια, που είναι και το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και τώρα παρακαλώ τον Επίτροπο να κάνει τον άθλο απαντώντας σε όλες τις παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλοι σας που κάνατε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ε, που ήταν συνήθως προς την ίδια κατεύθυνση. Χαίρομαι που κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή και ότι θεωρείται επίσης θετικό ε, να έχουμε φιλόδοξους εθνικούς ε, ολοκληρωμένους στόχους και σχέδια για το κλίμα και ότι χρειάζεται και ένα μακροπρόθεσμο όραμα για να ξέρουμε προς τα που οδεύουμε τα επόμενα χρόνια, διότι η κλιματική πολιτική δεν είναι κάτι που το συζητάμε μόνο μέχρι τι επόμενε εκλογέ. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρέπει να υπάρχει πολιτική συμφωνία μεταξύ χωρών, περιφερειών, δημών και κοινοτήτων για να πηγαίνουμε προ την ίδια κατεύθυνση. Μιλήσαμε για ενεργειακή απόδοση. Δεν αφορά ούτε τη δεξιότητα την αριστερά. Αφορά την ενέργεια, την ασφάλεια. Ε, να είναι φτηνότερο οι λογαριασμοί του ρεύματο για του πολίτε. Ε, πολλά είναι τα ωφέλη. Και σε αυτή την πολιτική απαιτείται καλή προετοιμασία και κατανόηση αλλά και δέσμευση, προσήλωση στους στόχους. Το μήνυμα λοιπόν που θέλω σήμερα να σας απευθύνω είναι πολύ ξεκάθαρο. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πραγματικότητα. 1,5 λέει το IPCC. Ήδη η θερμοκρασία έχει αυξηθεί έναν βαθμό ε, στην κλίμακα του Κελσίου από την προβιομηχανική εποχή και ανεβαίνει κάθε δεκαετία που σημαίνει τα επόμενα 50 ε, χρόνια ε, δεν θα καταφέρουμε από ό,τι φαίνεται να εφαρμόσουμε τους στόχους Παρίσιου με καταστροφικές επιπτώσεις για τον πλανήτη. Έξω και εμείς έχουμε τις πλέον φιλόδοξες συμβολές και όλους τους στόχους τους έχουμε εντάξει στην νομοθεσία και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Διότι οποιαδήποτε αλλαγή επισυμβεί στο πολιτικό πανόραμα, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, ο χάρτης, ο δικός, το φύλλο πορείας δεν αλλάζει, παραμένει το ίδιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όλοι δηλαδή να έχουν οικειοποιηθεί, όλες οι πλευρές να έχουν οικειοποιηθεί αυτά τα σχέδια. Κατά την εκπόνηση λοιπόν αυτών των σχεδίων θα πρέπει να ακούγεται η φωνή των δήμων κοινοτήτων, περιφερειών και να ακολουθούνται οι απόψει τους ε, και οι εισηγήσει τους. Ε. Γιατί αυτό ε, το έργο ξεκινάει στην πράξη επιτόπου, δηλαδή στο επίπεδο των Δήμων και Κοινοτήτων. Οι δήμαρχοι έχουν μεγάλο ρόλο, μίζωνα ρόλο πρέπει να οικειοποιηθούν, να έχουν την ιδιοκτησία των πολιτικών, να πείσουν δε και τους πολίτες, να τους μεταφέρουν τις αναγκαιότητες αυτές και να τους πείσουν πρέπει να προβούν σε αλλαγές για να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας και να μπορέσουν και αυτοί να συμμετέχουν στις συγκοινωνίες του αύριο και στην ενέργεια του αύριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος. Είμαστε στην πρώτη γραμμή. Δεν έχουμε εντελώς ε, καλύψει το ε, τους στόχους μας. Θέλουμε τη στρατηγική να την ε, ολοκληρώσουμε. Έχουμε όμως μια μακρόπνοη ε, εικόνα, ένα μακρόπνο όραμα. Ενεργειακή απόδοση θέλουμε να είναι στο επίκεντρο και σίγουρα η καλύτερη ενέργεια και η πιο καθαρή είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. 300 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο οργανισμό που πληρώνουμε ΣΥΟ ε, για τα ορυκτά καύσιμα. 400.000 ε, ε, Ευρωπαίοι πεθαίνουν πρόωρα λόγω κακής ποιότητας του αέρα, λόγω των εκπομπών και δίνουμε και επιδοτήσεις τουλάχιστον 40 δις. Λοιπόν, θα πρέπει να τα χωνέψουμε όλα αυτά. Αν δεν είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι, δεν θα μας ακολουθήσει κανείς. Είπα ε, είπαν θα φύγουν από τη Συμφωνία των Παρισιών. Η Κίνα που επενδύει πολύ σαν ανανόσιμες πηγές ενέργειας το 2030 θα φτάσει σε επίπεδο αιχμής. Εμείς θέλουμε να έχουμε μειώσει κατά 45% μέχρι τότε τις εκπομπές μας σε σχέση με το 99. Για όλα αυτά απαιτούνται επενδύσεις. Και εδώ έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που το αναφέρατε κι εσείς. Πρόκειται για τεράστια αλλαγή πολιτικής και δεν υπάρχει επιστροφή. Αλλάζει άρδινη κινητικότητα. Και αυτή η τεράστια αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς πολίτες. Αυτό είναι σαφές. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αν όλοι συμμετέχουμε και είμαστε έτσι προσιλωμένοι στην αλλαγή, ο αντίκτυπο αυτή τη μετάβασης δεν θα είναι ο ίδιος όλα τα εδάφη, γιατί υπάρχουν εδάφη που δεν θα ε, το καταλάβουν, ε, θα δουν τα ωφέλη μόνο, αλλά σε κάποια άλλα εδάφη που θα πρέπει να προσαρμοστούν εκεί θα χρειαστεί υποστήριξη. Σε ό,τι αφορά το λιγνί, το ρηκτά καύσιμα, το κάρβουνο, Θέλουμε να μειώσουμε τη συμβολή του στο ενεργειακό μείγμα και να αυξήσουμε το ποσοστό τη ανανεώσιμη ενέργεια. Έτσι όμω χρειάζεται υποστήριξη ε, στι περιοχέ αυτέ που θα βρεθούν σε μετάβαση. Επίση, ηλεκτροκίνηση ή κυψέλε υδρογόνου Πρέπει να υπάρξει πλήρη αναδιάρθρωση ολόκληρων περιφερειών, θα πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση ή απόκτηση νέων δεξιοτήτων για του εργαζομένου. Πρέπει να προετοιμαστούμε λοιπόν για αυτή τη μετάβαση, να διαθέσουμε και όλα τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να μην μείνει πίσω καμιά περιφέρεια. Και ταυτόχρονα πρέπει να πολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και στα σχέδια δράση ζητούμε από τι κυβερνήσει να αντιμετωπίσουν καλύτερα το πρόβλημα τη ενεργειακή φτώχεια. Και στι συστάσει ζητούμε να υπάρξουν διαβουλευσει με όλου του εμπλεκομένου φορείς. Άρα, μίζων ο ρόλο μα, σα ευχαριστώ και ε, εσά. Έχετε και εσεί, ίσω ακόμα πιο μείζον ρόλο να διαδραματίσετε. Γιατί εσεί είστε αυτοί οι οποίοι θα εφαρμόζετε επιτόπου αυτέ τι πολιτικέ. Δήμοι και κοινότητε και περιφέρειε ήδη είναι πιο φιλόδοξοι από ότι ε, ε οι εθνικέ κυβερνήσει στου στόχου που θέτουν. Αυτή τη διαδικασία πρέπει να την υποστηρίξουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάντοτε είναι μεγάλη χαρά μου να έρχομαι εδώ στην Επιτροπή των Περιφερειών και θα μελετήσω πολύ προσεκτικά και το τελικό κείμενο της γνωμοδότησής σας και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία και ελπίζω και στα επόμενα χρόνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα περάσουμε στην ιδέα τη τελευταία ε, γνωμοδότησης. Έχουμε καθυστέρηση βέβαια και πρέπει να επιταχύνουμε. Σα παρακαλώ να βοηθήσετε. Ο Εμιλιάνο, παρακαλώ. Εμιλιάνο, παρακαλώ. Ας έρθει γρήγορα εδώ.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 Monsieur le rapporteur, euh, vous avez la parole. Έχετε το λόγο κύριε Σίγητα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με συνέδρεμαν στην ε, κατάρτιση της έκθεσης. Πολλά πράγματα διδάχτηκα Η εμπειρία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πάνω απ' όλα αισθάνομαι περήφανο που Συντάσσοντα τη γνωμοδότηση, αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση, μπορέσα να εκπροσωπήσω την Επιτροπή των Περιφερειών και είναι η πρώτη μου εμπειρία αυτή. Θα ήθελα λοιπόν ιδιαίτερα να τονίσω τη σημασία τη παρουσίας και του τρόπου με τον οποίο μπορούν οι δήμοι και οι περιφέρειες να συμβάλλουν σε ένα δρόμο που δεν διστάζω να ορίσω ως ιστορικό για την Ευρώπη που θα οδηγήσει σε οικονομία ευημερίας, προόδου που δεν θα έχει συνέπειες αρνητικές στο κλίμα. Είναι πολλές λοιπόν οι ευθύνες μας, κοινέ οι ευθύνες, δεν αποκλείεται κανείς και με αυτό ως συνείδηση καταγράφω στην έκθεση τις προτάσεις, τις προτάσεις και τις δικές σας που ήταν πολύτιμες μέσα από ένα διάλογο πάρα πολύ ενδιαφέροντα και που επέτρεψε να ωφεληθώ και από τις δικές σας πολιτικές ιδέες και προτάσεις, πράγμα που δεν μου είχε συμβεί νωρίτερα. Χρειάζεται λοιπόν υγιείς πολιτικές η αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και αυτές πρέπει να χρηστούν από τη βάση προς τα πάνω. Όλοι συμφωνούμε πως πρέπει ο στόχος της αντιμετώπισης ε, ε, της κλιματικής αλλαγής και πάνω απ' όλα της συγκράτησης των συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας που μπορούν να την ε, επηρεάσουν στο 2050 είναι στόχος κοινό για τους Δήμους και τις κοινότητες. Καταγράφω με δυστημία του γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν κύρωσε αυτούς τους στόχους την προηγούμενη εβδομάδα με ομοφωνία. Το κείμενο της νομοδότησης ε, εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΕΝΒΗ με τις ε, τροπολογίες εκ των οποίων οι περισσότερες ε, τις οποίες και συμμερίζομαι έχουν βελτιώσει το κείμενο μόνο για ορισμένες χρειάστηκε να αντιπροτείνω τροπολογίες του εισηγητή συγκεκριμένα σε έξι, έξι τροπολογίες εισηγητή για να βελτιωθεί η διατύπωση να είναι πιο ευανάγνωστο το κείμενο θα σας τις παρουσιάσω πριν την ψηφοφορία δύο εκ των 33 τροπολογιών που έλαβα δεν μπόρεσα να υποστηρίξω, διότι θεωρώ πως αποδυναμώνουν το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα πρόκειται για την τροπολογία υπαριθμών 6 που έχουν προτείνει συντηρητική, ε, την οποία κρίνω απαράδεκτη καθώς ε, είναι σε αντίφαση με άλλες οδηγίες, με άλλες τροπολογίες που έχουν στο παρελθόν και άλλα κείμενα που έχουν στο παρελθόν εγκριθεί. Και αντίθετα με αυτό που προτείνει αυτή η οδηγία, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί ο δικό μα ρόλο σε αυτού του στόχου, στην επιτεύξη των στόχων αυτών και δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν οι επιδιώξει τη ε, εκθέσεω με μια τροπολογία όπω αυτή. Επίση, η παριθμόν 28, πάντα των συντηρητικών, περιγράφει ένα όραμα διαφορετικό από αυτό που προτείνει η έκθεση για το Carbon Capture Storage συγκράτηση και αποθήκευση άνθρακα. η οποία πιστεύουμε εμείς μπορεί να επιτευχθεί με τρόπους ε, φυσικούς όπως με το greening, όπως με την εξασφάλιση ε, φυσικών πόρων και δυνατοτήτων και μεθόδων ε, και όχι με την ε, αποθήκευση στο υπέδαφος του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή είναι, αυτές είναι οι δύο τροπολογίες και οι λόγοι τις οποίες, για τους οποίους δεν τις ενέκρινα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και προτείνω αμέσω να περάσουμε στη συζήτηση για τις τροπολογίες αυτές. Υπαριθμών 1 του εισηγητή αντικαθιστά την 1 και 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 3-4-5 ομού. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 7 του εισηγητή για να καταπέσουν οι 7, 8 και 9 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 του εισηγητή αντικαθιστά τι 10, 11, 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 και 14 ομού υπέρ κατά εγκρίνεται, εγκρίνονται 15 υπέρ κατά εγκρίνεται 16 του, του αντικαθιστά τις 16, 17, 18 αλλά με επιπλέον μια προφορική συμβιβαστική πρόταση τη βλέπετε στις οθόνες υπέρ Α, ζητάτε το λόγο. Με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει. Κύριε Λίμαν. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είμαστε κατά της τροπολογίας αυτής του εισηγητή και το υποστηρίζουμε τις 16 και 17 της κυρίας Ονέ και του κυρίου Κότς. Διότι αυτό που επιδιώκει ο εισηγητή είναι υπερβολικό σε όρου φορολογία. Χρειάζεται να υπάρχει κοινωνικά αποδεκτή φορολογία για να αποφεύγεται, παραδείγματι, το φαινόμενο που είδαμε στη Γαλλία ε, με τα κίτρινα γυναίκα. Πρέπει να δρούμε υπέρ και για του πολίτε, υπέρ των πολιτών και για του πολίτε και όχι εναντίον του. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Ποιο είναι υπέρ τη ε, τροπολογία του εισηγητή. κατά απορρίπτεται η τροπολογία αυτή οπότε πρέπει να ψηφίσουμε την κάθε τροπολογία ξεχωριστά τροπολογία 16 την αρχική 16 δηλαδή ψήφι ΠΕΡ. κατά εγκρίνεται τροπολογία 17 αρχική 17 ψήφι ΠΕΡ. κατά εγκρίνεται και Τροπολογία 18, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε ψηφοφορία, εγκρίνεται η 18. Προχωρούμε στην 19 τροπολογία του εισηγητού που αντικαθιστά τις 19, 20 και 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται τροπολογία 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται Έχουμε τώρα την τροπολογία 22, λέει ο συγητή, ο πρόεδρος. Α, συγγνώμη, έκανα λάθος, έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη. Τροπολογία 23, για την οποία υπάρχει προφορικός συμβιβασμό. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 25 του εισηγητού. Όχι, συγγνώμη. Μάλλον πηγαίνω λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Τροπολογία 24. Ψήφι περ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε το 25 του εισηγητή που αντικαθιστά την 25 έως 27 τροπολογίες Περ. Κατά εγκρίνεται. Επομένως πηγαίνουμε στο 28 ψηφιπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Le vote Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Η 28. Προχωρούμε στην τροπολογία 29 και προτείνω να ψηφιστεί από κοινού με τις υπόλοιπες και την 33. 29 33 αφού σας πω όμως ότι 31 έχει αποσυρθεί. Ψήφι υπέρ αυτού του μπλοκ τροπολογιών. Κατά εγκρίθηκε και περνούμε στην τελική ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Η γνωμοδότηση εγκρίνεται και συγχαίρω τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. τα σημεία 8 και 11 της ημέρας διάταξης που δεν θα μας απασχολήσουν πολύ θα καλοδεχθούμε, υποδεχθούμε τα νέα μέλη έχετε στο φάκελό σας ε, τις προτάσεις για τα νέα μέλη του Προεδρείου δεν βλέπω να έχει κασατήρηση να τους εγκρίνουμε ωραία εγκρίνονται η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει εδώ, στο ημικύκλιο, με την ακτήρια τελετή της 17ης εβδομάδας των πόλεων και περιφερειών και θα συνεχιστεί στις 8 και 9 στο κτίριο ε, Κάρλο Μάγνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπόλοιπες εργασίες μας. Και τώρα, σε μερικά λεπτά, θα έχουμε την κοινή τελετή που θα οργανώσουμε για την 25η επέτειο της ε, ε, ίδρυσής μας μαζί με το Κογκρέσο των Τοπικών και Ευρωπαϊκών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Chers collègues. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνοντα την ολομελιά μα, σα υπενθυμίζω ότι σήμερα συνεδριάζουμε για να συζητήσουμε τη διαδρομή ε, δύο οργανισμών που ασχολούνται με τις τοπικές και περιφερειακές ε, υποθέσεις δηλαδή του Κογκρέσου των τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου τη Ευρώπη και τη Επιτροπή των Περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι δύο οργανισμοί δημιουργήσαν εδώ και ένα τέταρτο αιώνα, το 1994, το πλαίσιο για αυτή τη συνεργασία. Έκτοτε σημειώσαμε μεγάλες επιτυχίες. Η συνεργασία μεταξύ των εργασιών ε, της Επιτροπής και του Κογκρέσου επέτρεψαν να υπάρξει περισσότερη αυτονομία και δημοκρατία στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να βελτιωθεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δημιουργήσαμε ε, μία κουλτούρα συνεργασίας, ένα κοινό όραμα. Κάθε φορά που χρειάστηκε να υπερασπιστούμε τις αρχές ε, που είναι τόσο σημαντικές ε, και για τους μεν και για τους δε. Επιδιώκοντας να αποφύγουμε τις επικαλύψεις όσο γίνεται, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να ακουστεί το σαφές μήνυμα των μεν και των δε, που βασίζεται στην ίδια αντίληψη για τις θεμελιώδεις αξίες μας. Το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η αποκέντρωση και την επικουρικότητα. Τα δύο θεσμικά μας όργανα επιδιώκουν πάντα να επιτύχουν τον καλύτερο συνδυασμό μεταξύ συμπληρωματικότητας και αποτελεσματικότητας για να έχουμε περισσότερη ε, επίδραση με λιγότερους πόρους. Είναι υπόδειγμα η συνεργασία μας γιατί έτσι υπερασπιζόμεθα τη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου συνολικά μέσω συγκεκριμένων δράσεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών επιτόπου που είναι η άμεση έκφραση αυτών των θεμελιωδών αρχών οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χρειάζεται και να ενισχύσουν τις ρίζες τους που είναι θεμελιώδης ιδρυτική αρχή τους αυτό που κάνουν μέσω του Κογκρέσου που επιτηρεί και δρά επιτόπου για να διασφαλίσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη σε βιώσιμη βάση. Αυτό γίνεται με βάση το πλαίσιο που ε, διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές της. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των, Θεμεριών, των Περιφερειών εγγυάται την εφαρμογή της επικουρικότητας. Η πολιτική συνοχής είναι καρπός ενός, μηχανισμού, ενός μηχανισμού άμεση συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Είναι βασικό θεμελιώδες εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και έχει υψηλή ορατότητα από τους πολίτες. Η άλλη πολιτική όπου συμβάλλουμε αποτελεσματικά είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων τις οποίες διαπιστώνουμε η πολυεπίπεδο διακυβέρνηση που προκύπτει από την κουλτούρα της αποκέντρωσης και της επικουρικότητας μας ε, οδηγεί σε ένα βασικό νομικό πλαίσιο όπου βασίζουμε την νομοποίησή μας η δημοκρατία και το κράτος δικαίου το Κογκρέσο και η Επιτροπή παρόλα αυτά έχουν πολύτιμα εργαλεία που πρέπει να αξιοποιηθούν για να ενισχύσουμε και να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου και την επικουρικότητα οι πρόσφατες ευρωεκλογές έστειλαν ένα θετικό μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία όσον αφορά τη συμμετοχή των συμπολιτών μας. Το επίπεδο συμμετοχής στις ευρωεκλογέ ήταν περίπου 51% για το σύνολο της Ένωσης. Ενώ το 2014 ήταν μόνο 43,4%. Προσωπικά όταν ακούω να αλληλοσυγχαιρόμεθα για το 51% ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το 49% που δεν ψήφισε σε πολλές χώρες οι ευρωεκλογέ έγιναν ε, παράλληλα με τοπικές, περιφερειακές ή ακόμη και εθνικές εκλογές όπως το Βέλγιο Αυτό ήταν θετικό γιατί κάνει την αναγκαία σύνδεση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Παράλληλα πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι η εμπιστοσύνη και η δέσμευση των πολιτών ποτέ δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Κατά συνέπεια, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να έχουμε την ίδια διαφανή προσέγγιση να αντιδρούμε στα ενάυσματα των πολιτών για να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και να αυξάνεται λοιπόν η ενεργό συμμετοχή τους. Μία από τις βασικές ε, αιτίες για τη δημιουργία μας το 1992 ήταν ε, η άνοδος της επιρροής ε, στην αρχή της δεκαετίας εκείνης των ευρωσκεπτικιστικών τάσεων. Θέλουμε να προσεγγίσει η Ευρώπη τους πολίτες διότι η Ευρώπη είναι πρώτα απ' όλα και κατά προτεραιότητα οι πολίτες της. Οι θεσμοί μας ήταν πάντα στο πλευρό των ε, δημάρχων και των τοπικά εκλεγμένων όταν υπερασπίζονταν τα καθημερινά δικαιώματα των πολιτών. Τα δικαιώματα που προκύπτουν από την πολιτική συνοχής η οποία επιτρέπει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να διαμορφώσουν το βιώσιμο μέλλον των περιοχών τους. Η Επιτροπή μας μας επιτρέπει επίσης να βγάλουμε ρίζες σε τοπικό επίπεδο. Χθε αναφερθήκαμε στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΠΑ. Τον περασμένο Απρίλιο συζητήσαμε τις πολιτικές ένταξης που ε, αναφέρονται στην Συμφωνία για τη Μετανάστευση. Για άλλη μια φορά, οι διεθνείς οργανισμοί, τα κράτη-μέλη, στρέφονται προς τοπικές και περιφερειακές αρχές όταν πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση. Επίσης, οι ε, νεαρές δημοκρατίες των Δυτικών Βαλκανίων βασίζονται στην αποκέντρωση και την επικουρικότητα για να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες τους οι οποίοι πολλέ φορέ ε, επαφίενται στου δημάρχου του για να ακουστεί η φωνή του ε, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών. Όλοι υπολογίζουν στι αρχέ τι δικέ μα για να γίνουν οι αναγκαίε μεταρρυθμίσει, για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, για να υπάρξει περισσότερη απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη. Συνοψίζοντα, η καλή διακυβέρνηση, η χρηστή διακυβέρνηση σε όλε τι μορφέ είναι προπόθεση για τη διατήρηση τη ελευθερία χαιρετίζουμε το θαυμάσιο έργο του Κογκρέσου, για παράδειγμα οι κανόνες διοντολογίας για όλους τους τοπικά και περιφερειακά εκλεγμένους. Είναι μόνο ένα παράδειγμα. Επίσης χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται τακτικά από το Κογκρέσο για να υπάρχει διαφάνεια και ανοιχτή κυβέρνηση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, μετά τις ε, συζητήσεις μας τώρα στις 2 η ώρα στην έδρα μας, στη, στο κτίριο Jacques Delors, θα έχουμε ένα σεμινάριο όπου θα συμμετέχουν ε, πολλοί μέλη του Κογκρέσου, όπου είστε όλοι προσκεκλημένοι. Και τώρα με πολύ χαρά να δώσω το λόγο στον συνάδελφο πρόεδρο του Κογκρέσου, τον Άντερς Κνάπε, που το γνωρίζουμε εμείς πολύ καλά. Ήταν συνάδελφός μας. Αγαπητέ Άντερς, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την θερμή υποδοχή. Χαίρομαι που είναι παρόντα τόσοι εκπρόσωποι και τη Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και του Συμβουλίου τη Ευρώπη σήμερα στο χαιρετισμό αυτό τη 25η επαιτίου. Είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι που μπορούμε να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση μαζί και σε πιο προσωπικό πνεύμα ως πρόεδρος ε, του Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλω να πω και λόγω του παρελθόντος μου στην Επιτροπή των Περιφερειών πως μεγάλη χαρά βλέπω αυτή την κοινή εκδήλωση. Χαιρετίζουμε λοιπόν μαζί σήμερα αυτήν την 25η επέτειο και όχι τυχαία γιατί είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους τα όργανα που εκπροσωπούμε και ε, έχει χάρη στην ε, συνεργασία μας βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων μας. Έχουμε μάλιστα την ίδια ηλικία ως ε, όργανα, πράγμα το οποίο δεν είναι και τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο γιατί η γέννηση των οργάνων που εκπροσωπούμε ε, συμπίπτει με μια συνειδητοποίηση της σημασίας των τοπικών και περιφερειακών αρχών και δομών στην Ευρώπη. Αρχικά είχε αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία διακρατικά και διακυβερνητικά μόνο. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφέ ότι πρέπει και η τοπική και περιφερειακή διάσταση να συμμετάσχουν, να συμπεριληφθούν στην ευρωπαϊκή συνεργασία και ολοκλήρωση. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην κοινοβουλευτική του συνέλευση ε, προσδίδεται μεγάλη σημασία και στην περιφερειακή και τοπική οργάνωση. Και έτσι λοιπόν το 1953 θεσπίζεται μια ειδική επιτροπή για τις περιφερειακές και τοπικές υποθέσεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το 1957 γίνεται και η πρώτη σύνοδος των τοπικών αρχών υπό την προεδρία του κυρίου Νταμά, Πρωθυπουργού τότε της Γαλλίας αλλά και Προέδρου μετά της ε, Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Και στη Βιέννη το 1993 εγκρίνεται η πρόταση για τη θέσπιση ενός συμβουλευτικού οργάνου που θα εκπροσωπεί, θα είναι ο γνήσιος εκπρόσωπος των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης, των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. από το 1957 έως το 1994 με την έγκριση των Υπουργών που θεσπίζει το Κογκρέσο στην φυσταμένη του μορφή ε, διαγράφεται μια μακρά πορεία ε, συνεργασίας μέσα από τις κεντρικές κυβερνήσεις και μέσα από ευρωπαϊκές δομές. Επίσης, χάρη στις πιέσεις από τις ε, περιφερειακές αρχές της, ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύεται στις ε, ευρωπαϊκές υποθέσεις η διάσταση της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης και έτσι στο Μάστριχτ έχουμε τη θέσπιση της Επιτροπής των Περιφερειών με εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Έτσι λοιπόν σημειώνουμε αυτή η σημαντική επέτειο από τη θέσπιση των δύο, θεσμικών, των δύο οργανών που εκπροσωπούμε ταυτόχρονα έχουμε συνολικά 70 χρόνια από την θέσπιση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επτά δεκαετίες αργότερα λοιπόν είναι σαφές πως ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη θεσμική δομή των κρατών μελών έχει όλο και πιο κρίσιμη σημασία. Έχει πιο κρίσιμη σημασία από ότι ποτέ η σημασία της δημοκρατίας είναι πλέον αναμφίβολη, επιτρέπει στον κάθε ε, πολίτη στην τοπική και περιφερειακή της διάσταση να αισθάνεται ότι μπορεί να ε, δρά, να συμμετέχει, να εκφράζει θέσεις και αξίες και να συμμετέχει βέβαια και στα όργανα από τον Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια, με μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μερικέ δεκαετίε και που έχει οδηγήσει σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα όπω άλλωστε αποδεικνύεται εσεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και εμεί, το Κογκρέσο Περιφερειών του Συμβουλίου τη Ευρώπη. με την έγκριση ενό ρυθμιστικού κειμένου του Ευρωπαϊκού Χάρτη τη τοπική αυτοκυβέρνηση. της τοπικής ε, ε, διακυβέρνησης και που τώρα έχει υιοθετηθεί από όλα τα κράτη ε, καταγράφεται η σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης ως χαρακτηριστικό κάθε δημοκρατικού καθεστώτος βέβαια πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε με χρυσό του αναγνωριστεί ο στην ουσία του ο κύριος ρόλος που διαδραματίζουν οι τοπικοί και οι περιφερειακοί εκπρόσωποι στις ε, δημοκρατίες μας. Εμείς ως Κογκρέσο των Περιφερειακών Αρχών σημειώνουμε με την ε, επιτήρηση των εξελίξεων σε ορισμένες περιπτώσεις ε, μια τάση των κεντρικών κυβερνήσεων να, ξανακέντρο, να ξαναοργανώνουν σε κεντρικό επίπεδο ή να διστάζουν ε, την παραχώρηση, την εκχώρηση τοπικές και περιφερειακές αρχές των πόρων που χρειάζονται για να επιτελέσουν το έργο τους. Και σε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα πρέπει να συνεχίσουμε με ιδιαίτερη έμφαση να προβάλλουμε τα, τις των τοπικών περιφερειακών αρχών και την παρουσία των εκπροσώπων τους. Ε, έτσι λοιπόν έχουμε κοινό αγώνα, υποστηρίζουμε τοπική δημοκρατία, τις δημόσιες πολιτικές στην Ευρώπη, ε, κάτω από την ίδια επιδίωξη κάτω από την ίδια παντιέρα χωρίς να έχουμε βέβαια το ίδιο δυναμικό και τις ίδιες δυνατότητες γιατί εσείς έχετε τις δυνατότητες που μπορεί να εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά οι δικές μας ως Συμβουλίο της Ευρώπης, ως Κογκρέσου Συμβουλίας της Ευρώπης είμαστε πολύ πιο περιορισμένοι στο Κογκρέσο όμως έχουμε την ε, δυνατότητα την προσπάθεια να χτίσουμε την τοπική δημοκρατία από τη βάση και προς τα άνω κάθε προσπάθεια γίνεται ε, βήμα το βήμα και από το χαμηλότερο επίπεδο προς το ανώτερο ενώ ναι, εσείς έχετε έχετε ρόλο να ε, παρέχετε συμβουλές με τις νομοδοτήσεις σας προς τα θεσμικά όργανα και βεβαίως ε, η ρόλη μας είναι διακριτή, ο καθένας μας το καθένα από τα δύο όργανα που εκπροσωπούμε ε, εργάζονται χωριστά, παράλληλα όμως και επιδιώκουν τον ίδιο στόχο, αυτό που ονομάζουν οι κυβερνήσεις επικουρικότητα μεν, εγώ όμως θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να αποκαλείται κοινή επιμερισμένη δημοκρατία. Έτσι λοιπόν ε, ο επιμερισμός της ε, διακυβέρνησης μεταξύ κεντρικής ε, κυβέρνησης και αποκεντρωμένων αρχών έχει μια διάσταση καθημερινού αγώνα, έχει μεγάλη σημασία και για το μέλλον της Ευρώπης πάντως και γνωρίζουμε σήμερα ότι μια συστοιχία απειλών κατά της Υπήρου μας που τις γνωρίζετε πολύ καλά αποτελούν και τη μεγαλύτερη πρόκληση που, αποτελεί Ευρωπαϊ... που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το τέλος Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και την ανάπτυξη της ε, πολυμερούς ε, συνεργασίας και των πολυμερών σχέσεων. Με το ε, Ευρωβαρόμετρο βλέπουμε ότι μόνο 36-38% των πολιτών αισθάνονται ακόμη εμπιστοσύνη επαρκή προς τις εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβουλιά τους, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνη των πολιτών μέχρι και 50 ή και πάνω από 40%. Πράγμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία σε μια εποχή διατάξης των ε, σχέσεων και της ισορροπίας και όταν γενικά η εμπιστοσύνη του πολίτη καταραίει προς τα όργανα που τον εκπροσωπούν έχει ακόμα μεγάλη εμπιστοσύνη ο πολίτης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και αυτές μπορούν να, το χτίσουν, να τον βοηθήσουν να χτίσει πιο γερές κοινωνίες. Είναι σημαντικές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δεν μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν πλέον σε ένα μονοδιάστατο επίπεδο. Υπάρχει ανάγκη για ευρεία ε, διαβούλευση, συντονισμένες ενέργειες, συμπληρωματικές δράσεις, συνέχεια στις επιλογές και στην πορεία από την τοπική μέχρι και την κεντρική εξουσία. Και πρέπει τα διαφορετικά επίπεδα της διακυβέρνησης να συνεργάζονται, καθώς ε, μόνο έτσι είναι δυνατόν να προχωρήσουμε οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, η τοπική και περιφερειακή δημοκρατία πρέπει πλέον να αναγνωριστεί ως ουσιώδης και εκ των ουκάνευ πυλώνας ε, των δημοκρατιών μας. η τοπική και περιφερειακή αιρετοί εκπρόσωποι είναι εκπρόσωποι των ε, πολιτών, των αρχών εκείνων που προσφέρει το κράτος στο επίπεδο το πιο κοντινό στον πολίτη και λέμε προς τις κεντρικές ε, κυβερνήσεις αξιοποιήστε αυτή την εγκύτητα που διαθέτουμε προς τον πολίτη κερδίστε και αυγατίστε αυτήν την εμπιστοσύνη που μπορεί να τρέφει ο πολίτης και αυτήν την ικανότητα να ε, πολλαπλασιάζει και να ενισχύει τη δημοκρατία η τοπική και η περιφερειακή αρχή. Εμείς εκπροσωπώντας τα δύο αυτά θεσμικά όργανα μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά ε, στην πορεία αυτή όπως άλλωστε έπραξαν τα όργανα που εκπροσωπούμε την τελευταία 25 ετία. Η επέτειος που εορτάζουμε σήμερα είναι ένας τρόπος να επενθυμίσουμε πως εμείς όπως και οι κεντρικές κυβερνήσεις έχουμε την ευθύνη της προαγωγής ενός σχεδίου για μια δημοκρατική Ευρώπη, για μια Ευρώπη ανοιχτή, για μια Ευρώπη που την ευήκονους προς τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ που μας προσφέρετε την ευκαιρία μέσα σήμερα να εορτάσουμε αυτή την επέτειο αγαπητοί συνάδελφοι και των δύο οργάνων Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα αυτό. Δράτω με της ευκαιρίας για να χαιρετήσω την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Κογκρέσου, Ανδρέας Φερισί, μαζί με τον Μπυριανέκ, το δικό μας Γενικό Γραμματέα, είναι από τους πυλώνες του στυλοβάτε της συνεργασίας αυτής ε, μεταξύ Συμβουλίου Ευρώπης ε, και Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής των Περιφερειών. Μια μακροχρόνια συνεργασία που σίγουρα θα έχει μπροστά της πολλές άλλες προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Και φτάνουμε στο σημείο που θα ακούσουμε παρεμβάσεις από εσάς καθώς και από μέλη του Κογκρέσου. Έχουμε κάπως αναμίξει τη σειρά, να υπάρχει μια ισορροπία. Η Ευρώπη θέλουμε να είναι ισορροπημένη άλλωστε. Και ισορροπή εκπροσώπηση των δύο φίλων λίγο πολύ βλέπω. Με απόδειξη απτή το ότι η Ελένη Λουκαίδου είναι η πρώτη ομιλήτρα που θα πάρει το λόγο. Merci. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Άντερς, αγαπητέ Καρλ Χάιντς, ε, είναι τιμή ε, και χαρά μου να απευθύνω ε, με σε εσάς εκ μέρους όλων των μελών του ΕΛΚΑ από την Επιτροπή των Περιφερειών προς εσάς όχι μόνο γιατί είστε ένας φίλος από τα παλιά, αλλά και γιατί είστε ένας στρατευμένος φίλος στο πλαίσιο του ΕΛΚ για πάνω από 20 χρόνια και η Επιτροπή των Περιφέρων και το Κογκρέσο εργάζονται για να προωθήσουν τα συμφέροντα ε, των λαών, για τους λαούς, για να ενισχύσουν τα θεμέλια μιας κοινή ιδέας. Δημοκρατική, δηλαδή δίκαιη και ευημερούσα Ευρώπη. Και αυτή η Ευρώπη ξεκινάει από τα χωριά, από τις πόλεις και από τις περιφερειές μας. Εξού και πρόκειται για κοινό χρέος, κοινό καθήκον. Να ακούσουμε, να αφογκραστούμε τον κόσμο στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο και την φωνή του να την μεταφέρουμε στο επίκεντρο, στην καρδιά της ευρωπαϊκής συζήτησης. Από κοινού μπορούμε να συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας Ευρώπης που θα προστατεύει τους πολίτες της και θα τους κάνει πιο χαρούμενους, πιο ευτυχισμένους. Και θεωρώ ότι η επέτειος που γιορτάζουμε σήμερα είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία για να αναστοχαστούμε το μέλλον της Ευρώπης, οπότε ολοκληρώνοντας θέλω να σας πω ότι φέτος δεν ότι μόνο αυτή η χρονιά, την 25η επέτειο τη συνεργασίας μεταξύ Επιτροπή Περιφέρειων και Κογκρέσου, αλλά είναι και μια χρονιά κρίσιμων αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης, το δικό μας το μέλλον. Το ΕΛΚΑ σας ενθαρρύνει και ε, θέλουμε να είμαστε όλοι ενωμένοι, να σταθούμε μαζί σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς ατενίζοντας ένα μέλλον που θα ε, λαμβάνει υπόψη και θα σέβεται τις προσδοκίες των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. από το συνέδριο τώρα, το Κογκρέσο επόμενος ο μιλητής ε, Präsidenten, Αξιότιμοι πρόεδροι, αξιότιμοι συνάδελφοι, συγχαρητήρια σε αυτή την κοινή επέτειο, συγχαρητήρια και στο Προεδρείο που έλαβε την πρωτοβουλία για την ε, ε, κοινή αυτή τελετή εορτασμού της επέτειου Πολλά πετύχαμε φέτος, σίγουρα όμως παραμένουν πολλά σημαντικά επιτεύγματα να πετύχουμε. Έχουμε αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό, τα έχουμε πει, υπάρχουν κάποιες νέες τάσεις ε, συγκέντρωσης, ενώ εμείς θέλουμε αποκέντρωση. ενώ βλέπουμε τάσεις συγκέντρωσης ε, είτε οθούμενης από πολιτικούς λόγους είτε από οικονομικούς. Σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εμείς έχουμε την μοναδική ευκαιρία να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες οι οποίοι μας περιβάλλουν με εμπιστοσύνη εμάς ε, τους ε, τοπικούς περιφερειακούς ερετούς και αυτό είναι μια ευκαιρία για τη δημοκρατία γιατί ε, βλέπουμε να μειώνεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και εμείς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση και να ενισχύσουμε το τοπικό περιφερειακό επίπεδο και θα πρέπει να ενισχύσουμε την τοπική δημοκρατία. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, παραδείγματο ψηφιοποίηση, πώς λειτουργεί σήμερα ο διάλογος με τους πολίτες, ψηφιοποίηση κοινωνικά μέσα δικτύως και πολλά άλλα θέματα. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι πολίτες ε, σε αυτό το επίπεδο. Άλλα θέματα σημαντικά είναι χάρη η προστασία του κλίματος, στόχη της βιωσιμότητας και στο τοπικό επίπεδο μπορούμε από κοινού να προωθήσουμε αυτούς τους στόχους. Ε, θα ήθελα λοιπόν και προσβλέπω ε, στη συνέχιση της εργασίας αυτής εμείς από το ΕΛΚ είμαστε φυσικά στην πρώτη γραμμή. Ας προχωρήσουμε, ας δουλέψουμε όλοι για την ενίσχυση τοπικής περιφερειακής δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπίργκιτ Χονέ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Αξιότιμοι κύριοι πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου στα συγχαρητήρια για τα 25 χρόνια συνεργασίας μεταξύ των ε, Δήμων Κοινοτήτων, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής Περιφερειών και Κογκρέας Τοπικών Περιφερειακών 25 χρόνια μεγαλύτερης ολοκλήρωσης, μιας μεγαλύτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμβάλλουμε κι εμείς στη συνοχή της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι από την ε, Σαξονία. Εμείς ε, και στις δύο οργανώσεις ε, συμμετέχουμε ενεργά και χαιρετούμε, χαιρετίζουμε αυτή την συνέργεια μεταξύ της ε, τη Επιτροπή των Περιφερειών και του Κογκρέσου και θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο για να ενισχύσει την τοπική και περιφερειακή δημοκρατία στην Ευρώπη. Αυτή η επέτειο πρέπει να αξιοποιηθεί, να είναι μια ευκαιρία να ταινίσουμε την επόμενη 25 αιτία που είναι μπροστά μα. Τι είναι τα βασικά, οι βασικέ προκλήσει. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να έχουμε επιτυχή πολιτική συνοχή που θα πρέπει να είναι η βάση για ε, συνέχιση αυτή τη κοινή ανάπτυξη και βελτίωση εξέλιξη Ένωση. Δεύτερον, θέλουμε φιλόδοξη προστασία του κλίματο με μια βιομηχανική πολιτική που θα είναι καινοτόμο, ε, που θα την προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα την εφαρμόζουν στην πράξη οι ε, Δήμοι και οι Περιφέρειε. Τρίτον, θέλουμε κοινωνικό πυλώνα πιο ισχυρό ε, και πρωτοστάτη την, την Επιτροπή των Περιφερειών για τη συνοχή της κοινωνίας και θεμέλιο ε, μιας επιτυχημένης δημοκρατικής κοινωνίας. Τέταρτον, θέλουμε Επιτροπή των Περιφερειών ε, που θα έχει πιο ενεργό ρόλο στον όλο πολιτικό κύκλο και στις δικασίες λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή των Περιφερειών, κυρίες και κύριοι, μας φαίνει πιο κοντά στην Στου Δήμους και τις Περιφέρειες και εμεί εμείς φέρνουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους Δήμου και τις Περιφέρειες πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πολύ σημαντικό και στηρίζω επίσης ε, το διάλογο των πολιτών ε, ώστε να καταστεί μια μόνιμη δομή. Ε, αυτό πιστεύω ότι θα ενισχύσει την τοπική περιφερειακή δημοκρατία και τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη εν γέννη. Μόνο θετικά ωφέλη μπορώ να προκύψουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Φασίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον, τον Πρόεδρο Λάμπερτ, να τον ευχαριστώ για την πρωτοβουλία αυτή και ιδιαίτερα να απευθύνω χαιρετισμό προ τη σοσιαλιστική ομάδα του Κογκρέσου των Οπικών και Περιφερειακών Ορχών του Συμβουλίου τη Ευρώπη και όλου του εκπροσώπου που βρίσκονται εδώ, εκ μέρου μάλλον του Συμβουλίου. Και αν θέλει ένα πολίτη για οποιοδήποτε λόγο να βρει λύση σε ένα πρόβλημά του, θα πάει στον Δήμαρχο, θα πάει στι τοπική ε, αρχέ, στις αρχές που είναι και η πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των αγκών του πολίτη. Ε, μια οικογένεια με μικρά παιδιά που χρειάζεται φερρυπίν παιδικό σταθμό ή άλλες τις υπηρεσίες θα πάει στο Δήμαρχο. Ένας πολίτης που έχει μέλημα για το περιβάλλον και την καθαρή ατμοσφαιρική, την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα το ίδιο θα πράξει. Όποιος έχει επαγγελματική εμπορική δραστηριότητα και χρειάζεται στηρίξη θα πάει στο τοπικές, στις δημοτικές του αρχές. Ε, όποιος επιδιώκει να προχωρήσουν ε, ε, οι υποδομές σε μια περιοχή να είναι πιο καλές οι μεταφορές θα στραφεί προς τις αρμόδιες ε, αρχές της τοπικής ε, αυτοδιοίκησης. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα που να αφορά την καθημερινή ζωή των οικογενειών που να περνά από το γραφείο των τοπικών αρχών. Ακόμα και τα θέματα τη μετανάστευση περνούν μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν θεωρεί κάποιο ότι μπορεί να ζει ε, σε μια περιοχή, σε έναν δρόμο που δεν είναι αρκετά ασφαλή, θα πάει στην αστυνομία. Και καλείται τώρα ο ένα δήμαρχος να αγγιηθεί και την ασφάλεια των πολιτών. Και έτσι νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο καθώ ε, οι τοπικές αρχές έχουν ε, κληθεί πλέον να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στις προσδοκίες των πολιτών και είναι αυτή η τοπική δημοκρατία ο θεμελιώδης πυλώνας για την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει ο πολίτης στην πολιτική. Μια στιγμή χρονική, μια περίοδο χρονική όπου είναι μεγάλη η δυσπιστία για να μην πω η εχθρότητα εναντί των ε, δομών της πολιτικής. Οι τοπικές αρχές είναι ένας απαραίτητος ε, κρίκος, μια γέφυρα που μπορεί να επιτρέψει να να ξαναχτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη αρκεί να είναι ισχυρές βεβαίω και αυτό είναι ο αγώνα μα, για ταυτόχρονα ε, είναι αγώνας για την ενίσχυση της δημοκρατίας γι' αυτό εργάζεται και το Κογκρέσο των Οπικών Αρχών και η Επίτροπη των Περιφερειών γι' αυτό και πρέπει να εορτάζουμε τι 25 χρόνια ε, ύπαρξης και συνεργασία και βεβαίω να προσβλέπουμε στην επόμενη 25 ετία Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Μπουκάναν Ευχαριστώ. Και σας συγχαίρω και τους δύο ε, και τις οργανώσεις σας. Λέγομαι Τόνι Μουκάναν. Είμαι από τη Σκωτία, επικεφαλής μιας κομιτείας και είμαι μέλος και των δύο οργανισμών. Ε, νομίζω ότι είμαι ο μόνος, ίσως, ε, αλλά σίγουρα είμαι ο μόνος από τη Σκωτία. Έχω δει και τις διαφορές και τις ομοιότητες των δύο οργανισμών, των δύο φορέων. Και εγώ και οι συνάδελφοι από τη Σκωτία έχουμε υπάρξει συγκητές ε, στους διάφορους ε, και στους δύο θεσμούς. Ο κύριος Μακουίγκαν ήταν εισηγητής για μια έκθεση για τις αλλαγές στην τοπική δημοκρατία στην Ευρώπη. Ο κύριος Οχέρν πολύ πρόσφατα έκανε μια έκθεση του Κογκρέσου για την ε, δημοσιονομική αυτονομία του Κογκρέσου. Και εγώ Είμαι, έχω υπάρξει συζητητής και για θέματα γεωργίας και για θέματα αλίας και έχω εκπροσωπήσει το Κογκρέσο στη συνάντηση κορυφής για τη διαφάνεια και για, σε μία άλλη εκδήλωση για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Από αυτή την ε, άποψη, εάν ε, τελικά γίνει Brexit και αν δεν είμαστε σε θέση να συμμετάσχουμε, και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το κάνουμε ως ανεξάρτητο έθνος. Θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Θέλουμε να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα επαφής μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Επιτροπής των Περιφερειών για να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ευρώπη και την περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κόλτς Κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε. Η δημοκρατία είναι άρρωστη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σε διάφορα μέρη, σχεδόν παντού, βλέπουμε να ε, ανεβαίνει η επιρροή λαϊκιστικών κινημάτων της ακροδεξιάς ή της, εκρο... της ακροαριστεράς. Ε, υπάρχουν πολλά αίτια. Δεν προλαβαίνω να τα αναφέρω, αλλά η πεποίθησή μου είναι. Είναι ότι για να ενθουσιαστεί και πάλι ο συμπολίτη μας για την πολιτική Πρέπει να περάσουμε από το, νομικό, από το τοπικό επίπεδο. Η δημοκρατία είναι ένα κεκτημένο για το οποίο πρέπει πάντα να αγωνιζόμαστε. Η δημοκρατία δεν δημιουργείται μόνο από τα πάνω, αλλά και από τα κάτω. Και θα έλεγα πρώτα απ' όλα από τα κάτω. Γι' αυτό η εγκύτητα που είναι ο Δήμος και η κοινότητα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να τα υπερασπιστούμε, να τα προωθήσουμε. Αυτή είναι η έννοια της συμπληρωματικότητας ε, της δράσης των δύο θεσμών μας, την οποία εορτάζουμε σήμερα. οι ε, τοπικοί και οι περιφερειακά εκλεγμένοι είναι πραγματικά οι καλύτεροι εκλεγμένοι. Είναι συναρπαστικό να είσαι σε άμεση επαφή με τους ε, συμπολίτες σου και να μπορείς να επηρεάζεις την ε, εξέλιξη των πραγμάτων στη γειτονιά σου. Σε αυτό το επίπεδο είναι ζωντανή δημοκρατία και ο πολίτης μπορεί να εμπλακεί περισσότερο σε επιλογές που τον αφορούν. Πρέπει να το επενθυμίζουμε συνεχώς στις κυβερνήσεις μας. Γιατί πολύ συχνά ενδίδουν στον πειρασμό της, ε, του συγκεντρωτισμού. Εμείς επιδιώκουμε το αντίθετο. Χαίρομαι που όλοι μας δεσμευόμεθα για την τοπική και περιφερειακή αυτονομία, αλλά δεν αρκεί απλώς να το τονίζουμε. Πρέπει επίσης να κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει οι οργανώσεις μας να ιδρώσουν τη φανέλα, να κάνουν περισσότερα, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η αυτονομία, γιατί σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιοχές Υπάρχει τάση ε, συγκεντρωτισμού, επαναφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων σε κεντρικό επίπεδο. Άρα πολλά έχουμε ακόμη να κάνουμε και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. David Simmons. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ίσως ε, ε, είμαστε αρκετοί που είμαστε μέλη και των δύο οργανισμών που μιλάμε. Από πλευρά του ECR λοιπόν θέλω να αναφερθώ και εγώ στο πόσο θετική είναι αυτή η επέτειος. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι είμαστε οι δύο πυλώνες της, ε, ότι, συγγνώμη, οι δύο πυλώνες ε, της δημοκρατίας μας είναι το κράτος δικαίου και η δημοκρατία. Και η Επιτροπή των Περιφερειών εκπροσωπούν τη δημοκρατία ενώ εμείς ε, και γενικά το Συμβούλιο της Ευρώπης εμείς ως Κογκρέσο δηλαδή εκπροσωπούμε το κράτος δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές οι δύο θεσμοί γιατί ναι μεν διαφορετικός ο ρόλος μας αλλά η δυνατότητα και ε, το προσωπικό μας και εμείς οι ίδιοι να ανταλλάσσουμε απόψεις για το πώς αντιμετωπίσαν προκλήσεις ε, είναι ανεκτήμητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο πιστεύω του τρόπου με τον οποίο συνεργαζόμαστε παντού στην Ευρώπη. Όχι μόνο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ευρύτερα. Όλα τα ευρωπαϊκά έθνη. Και καταλήγοντα. Δύο κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικά σημεία. Πρώτον, στη σημερινή πολιτική συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε τη διατήρηση του σεβασμού για την αλήθεια και για την ε, δέουσα διαδικασία που υφίστανται πολλέ πιέσει και βεβαίω στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε δέσμευσή μα προ αυτή την κατεύθυνση. Όλοι μα που είμαστε πολιτικοί των κυρίων κομμάτων πρέπει να θέσουμε κατά μέρο τι διαφορέ μα που είναι κατανοητέ, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι είμαστε και πάλι σε επαφή με του ψηφοφόρου μα, ούτω ώστε να κατανοήσουν ότι τα κύρια κόμματα ασχολούνται με τα συμφέροντά του, την ευημερία του και εργάζονται επιμελώ για θέματα που του αφορούν. Και δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε σαφή καθορισμό προτεραιοτήτων. Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι ανησυχούν ότι η κατάσταση, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, όσον αφορά τη συνεργασία για την παρατήρηση των εκλογών, παρεμποδίζεται από την έλλειψη χρηματοδότηση. από πλευρά τη ομάδα μου, του ECR. Κάνω έκκληση να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την πολύτιμη δουλειά για να βοηθήσουμε όλου του συναδέλφου που χρειάζονται τη δημοκρατία από όπου και αν προέρχονται. Ευχαριστώ

Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό, θα ξεκινήσουμε αμέσω. Ladies and gentlemen, on the 25th anniversary of the Congress of Local and Regional Authorities. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με την 25η αυτή επέτειο του Κογκρέσου θα ήθελα να σας καλωσορίσω ε, όλους και να χαιρετήσω αυτή την επέτειο. Соціальна справедливість невід'ємні від економічної свободи, і ми активно відстоїмо ці принципи. Ως μέλος ιδρυτικό της πολιτικής μας ομάδας θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έφαση στο γεγονός πως δίνουμε μεγάλη σημασία στην πολιτική ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη ε, που είναι αναπόσπαστα δεδομένα την οικονομική ελευθερία. Το Κογκρέσο και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι στρατηγικοί εταίροι και μπορούν να προβάλλουν από κοινού το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών και να ε, το Συμβούλιο των Υπουργών για να συζητήσουν κέρια θέματα. Uh, Εκπροσωπούμε διαφορετικές χώρες, διαφορετικές οργανώσεις, ταυτόχρονα όμως είμαστε η μία φωνή των τοπικών αρχών στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και χαιρόμαστε που μπορεί να ακουστεί αυτή η φωνή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από τα σύνορά της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 αποδεικνύουν πως παραβιάζονται οι αρχές και οι αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και βέβαια ότι γίνεται εκβιασμός οικονομικός και άλλος από την Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι συμβολική το ότι ακούγεται σήμερα η Ουκρανική γλώσσα σήμερα είναι και μια ένδειξη σεβασμού για μας. Демократію, свободи і принципи Європейської хартії місцевого самоврядування. Довіра до наших інституцій не має ставитись під сумнів за будь-яких умов. Дякую. We must be united in... Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, προστατεύουμε τη δημοκρατία, τις ελευθερίες, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν πρέπει ποτέ να φημώνεται αυτή η φωνή. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ και θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, Επιτροπή των Περιφερειών και το Κογκρέσο για τη μεγάλη αυτή επέτειο έχουν καταστεί και τα δύο όργανα αυτά πολύ χρήσιμα εργαλεία για την προαγωγή της τοπικής και περιφερειακής ε, αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη. Πάντοτε η καταλανική κυβέρνηση θα αγωνίζεται για την προαγωγή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε υπέρ της Ομοσπονδιακής Ευρώπης. Θεωρούμε ότι είναι ο μόνος τρόπος να βελτιωθούν οι ζωέ των ανθρώπων. Η επιλογή τη ομοσπονδιακή Οργάνωσης σημαίνει ότι και ξεφεύγουμε από το, τη λέσχη των μεγάλων κρατών που έχει φανεί να ε, απεικονίζει την Ευρώπη αλλά και ταυτόχρονα ερχόμαστε πιο κοντά στο επίπεδο του πολίτη και προσβληθούμε στη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και το Κογκρέσιο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την ενίκηση του έργου, για την προαγωγή της ποικιλία και όλων των δημοκρατικών δυνάμεων στα ευρωπαϊκά εδάφη. Le prochain orateur est Peter Florian Schütz. Πέτερ Φλόριαν Σούτς, επόμενος ομιλητής. Αξιότιμοι πρόεδροι, αξιότιμοι συνάδελφοι, μια ωραία μέρα ζούμε σήμερα. Γιορτάζουμε αυτή την επέτειο που Ουσιαστικά ε, είδαμε να δημιουργείται η Ευρώπη επιτόπου σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Μια Ευρώπη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και έχουμε και τον αδελφό μας ε, εδώ οργανισμό, το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, με τον οποίο εκπροσωπούμε από κοινού τις ίδιες αρχές, ανθρώπινα δικαιώματα, ασφάλεια, κράτος δικαίου και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό και γι' αυτό το οποίο πετύχαμε τα τελευταία 25 χρόνια γιατί δείχναμε ότι εφαρμόζουμε στην πράξη τις αρχές αυτές και το ίδιο ελπίζω να γίνει και στις, στην επόμενη 25 ετία και στη χώρα μου και στην πόλη μου ε, την ε, Βιέννη ε, κάνουμε πολλά το θέμα είναι ότι πρέπει να Λάβουμε υπόψη ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η Ευρώπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τώρα λέει ο πρόεδρος είναι το λόγο στον συνάδελφο Καλαμπουίκ. Ευχαριστώ πολύ και στους δύο πρόεδρους. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη δουλειά που έχετε κάνει. Γιατί ο ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών είναι αυξανόμενος. Αυξάνει το γόητρο, η επιρροή, η συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών στην ορατότητα, στην προβολή και τη σημασία των περιφερειών για τη συνδιαμόρφωση του συνόλου Ένωσης. Θέλω να επιμείνω ε, στο ότι δήμοι και περιφέρειες είναι οι θεσμοί ε, που χαίρουν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών. Άρα είναι κάτι πολύ θετικό. Ε, και ακούω και περισσότερο η Ένωση, την Επιτροπή των Περιφερειών και αυτό πρέπει να συνεχίσει να πράττει. Είναι μια σωστή συνετή προσέγγιση. Ο διάλογος των πολιτών, γιατί εμεί είμαστε κοντά στου πολίτες, είναι ένα διάλογο που πρέπει να γίνεται συνεχώ. Επίσης, να γίνεται στο πλαίσιο πλαίσιο των αρχών που συμμεριζόμαστε και κράτος δικαίου, ε, δικαιοσύνη, ελευθερία. Το κράτος δικαίου είναι κάτι πολύ σημαντικό ε, γιατί εμείς είμαστε σημαντικοί γιατί εφαρμόζουμε τις πολιτικές δράσεις, τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και ιδίως στο κοινωνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής. Μάικ η 20η και 25η σε σημαντικά, ε, σε, σημαντικές επέτειοι πρώτη ε, από το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου και η δεύτερη αυτή τη ε, συνεργασία. Εγώ τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είχα την τιμή να συμμετάσχω ε, και στο ε, προσπάθεια ενίσχυσης της Ουκρανίας που είναι στο δρόμο του εκδημοκρατισμού και με την Επιτροπή των Περιφερειών ήμασταν στο Μαϊντάν για την Ουκρανική Επανάσταση αλλά και μετά ήμασταν εκεί. Παρακολουθήσαμε τι κάνει η Ουκρανία με τους Δήμους, τα Δημοτικά Συμβούλια και χαιρετήσαμε την πορεία εκδημοκρατισμού της Ουκρανίας. Κάτι πρέπει να συνεχιστεί. Το είδαμε, είδαμε την αξία ε, και με την Task Force ε, τη επιτροπή μα. Όμως ε, θέλω να σχολιάσω αυτά που είπε νωρίτερα εκπρόσωπο. Η πρόσφατη απόφαση της κοινοβουλευτικής συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη να ξαναδεχθεί τους εκπροσώπου της Ρωσική Ομοσπονδίας μερικοί είναι και από την κατεχόμενη Κρυμαία. Όταν Βλέπουμε ε, ε, ακόμα ε, τα συντήματα του M16 το οποίο και υπονομεύεται η δημοκρατία εκεί και από τη Ρωσική Ομοσπονδία όλα αυτά ε, υπαγορεύονται. Αυτά υπονομεύουν την πολύ καλή δουλειά που έχουμε κάνει εμείς μέχρι τώρα και νομίζω ότι σε αυτήν την επέτειο πραγματικά είναι επέσχυντο να έχουν γίνει τέτοια αρνητικά ε, συμβάντα. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε ως Επιτροπή των Περιφερειών να βρισκόμαστε στο πλευρό των Ουκρανών στο δρόμο προς τη μετάβαση και τον εκδημοκρατισμό. Ευχαριστώ πολύ όλους τους Και τώρα παρακαλώ τον Άντα Κνάπε να κάνει μια ολοκλήρωση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολλά από τα θέματα που θήκησαν κατά συζήτηση. επηρεάζουν ε, την τοπική διακυβέρνηση όλα τα 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης άρα και όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διορθώσει κάποιες ε, αδυναμίες. Ε, πρέπει να υπάρχει επίσημη διαβούλευση μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικών και περιφερειακών αρχών για θέματα που αφορούν τις τελευταίες. Όχι μόνο οικονομικής φύσης, αλλά οποιοδήποτε θέμα που έχει να κάνει με τι αρμοδιότητε και τα καθήκοντά του και τη δυνατότητα να έχουν αυτά αποτελέσματα για του πολίτε του. Αυτά τα βλέπουμε μέσω των ε, διαδικασιών επιτήρησης που κάνουμε. Διαπιστώνουμε ότι οι τάσεις είναι αρνητικές. Πολύ συχνότερα οι κεντρικέ κυβερνήσει παίρνουν αποφάσεις παρά το ότι γνωρίζουν, το παραβιάζουν αυτά τα οποία έχουν υπογράψει στην Σύμβαση για την τοπική και περιφερειακή δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και η Επιτροπή Περιφερειών όταν συζητά τη σχέση με την κεντρική κυβέρνηση να αναφέρεται σε αυτήν την χάρτα. Πρέπει λοιπόν για αυτό το θέμα να εργαστούμε ενωμένοι. για να διορθωθεί η κατάσταση. Να τηρούν τη χάρτα την οποία υπέγραψαν τα κράτη-μέλη. Αλλά όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχουν και πολλά άλλα κοινά συμφέροντα. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Έχουμε την κατάσταση της μετανάστευσης. Το θέμα της μετανάστευσης. Το δημογραφικό θέμα βλέπουμε ότι ο πληθυσμός μας είναι όλο και γυρεότερος με όλες τις επιπτώσεις είναι πολύ θετικό το ότι ζούμε περισσότερο, ότι είμαστε ευπορότεροι, υγιέστεροι. Αλλά αυτό ασκεί πίεση επί των τοπικών και περιφερειακών αρχών που πολύ συχνά είναι υπεύθυνε για πολλούς τομείς ε, της αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή Περιφερειών και για το Κογκρέσο μας είναι ε, η αυξανόμενη διαφθορά που είναι δηλητήριο για τις κοινωνίες μας. Δημιουργεί δυσπιστία έναντι των ε, εκλεγμένων εκπροσώπων σε κάθε επίπεδο. Πρέπει να εντείνουμε την καταπολέμηση διαφθοράς και οι δύο μας θεσμοί. Επίσης υπάρχουν ε, απειλές κατά των ε, ηγετών μας, των εκλεγμένων ηγετών μας, παντού στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο απειλέ από κάποιους ε, μεμονωμένους πολίτες, αλλά και από διάφορες ε, εγκληματικές συμμορίες και από άλλους πολιτικούς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Διότι αυτό σημαίνει ότι πολλοί αποφεύγουν ε, να ε, μπουν σε ψηφοδέλτιο ή να ασκήσουν καθήκοντα εκλεγμένου γιατί είναι πολύ ε, αξιόπιστες και βαριές αυτές οι απειλές. Επίσης, το θέμα ισότητας φύλων πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Υπάρχουν πολύ σαφείς κανόνες στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ότι κάποιο φύλλο υποεκπροσωπείται και θέλουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση να εκπροσωπούνται εξίσου και τα δύο φύλλα. Και όπου έχουμε επιτύχει να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά το θέμα αυτό, τότε διαπιστώσαμε κατόπιν ότι αυξήθηκε η αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Τέλος. Ως Κογκρέσο είμαστε ανοιχτοί και προσβλέπουμε ότι στα επόμενα 25 χρόνια θα υπάρξει ένταση της συνεργασίας μας γιατί είμαστε αλληλοσυμπληρούμενοι. Σας διαβεβαιώ κύριε Πρόεδρε ότι από πλευρά Συμβουλίου της Ευρώπης είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε. Ως Κογκρέσο δεν μας χαροποιεί η κατάσταση όπως είναι τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσον αφορά την εκπροσώπηση και τις αποφάσεις που λήφθησαν. Και ξέρω ότι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι συμφωνούν. Υπονομεύεται έτσι η αξιοπιστία ενός θεσμού που έχει τρεις στόχους. Δημοκρατία, κράτος δικαίου και Θα συνεχίσουμε ως Κογκρέσο να, συνεχ... να συζητάμε με τους φίλους από τις τοπικές αρχές και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες γιατί η κατάσταση όπως έχει τώρα είναι απαράδεκτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ε, καταληκτικές σας παρατηρήσεις που καταδεικνύουν ε, δυνατότητες συνεργασίας. Θα συνεχίσουμε την κοινή μας ε, εξέταση των θεμάτων αυτών από τις 2 και μετά στο κτίριο Jacques Delors της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφυρών στην αίθουσα 52 όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την κατάσταση της αποκέντρωσης στην Ευρώπη. Αλλά πριν από αυτό πρέπει όλοι κάπως να ε, ε, ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας. Οπότε σας καλώ στο πέμπτο όροφο στο έθριο που έχουμε εκεί όπου θα έχουμε ένα περιπατητικό γεύμα θα έχουμε δυνατότητα βέβαια ε, να πούμε περισσότερα άρα δεν ξέρω θα προλάβουμε να φάμε γιατί όσο περισσότερο μιλάς τόσο λιγότερο τρως ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας ελπίζω να τα ξαναπούμε αλλά σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι εξαίρετες διακοπές και να επανέλθετε πλήρης δυνάμεων για να κάνουμε την τελευταία ευθεία της θητείας μας στις Ολομέλειες του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου ως Επιτροπή Περιφερειών και ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι όλα τα προβλήματα της Ευρώπης να επιληθούν ως διαμαγείας. Σας ευχαριστώ πολύ.